Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες μας και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουμε μια ανακοίνωση του κυρίου Γιώργη Νίγες Φερέρ που ήρθε για να παρουσιάσει τις εργασίες που έγιναν περί των τρόπων ε, καταλογισμού στους εθνικούς προπολογισμού των συμμετοχών στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2014 ένα παλιό μέλος της Επιτροπής μας, ο Ζαλιγκδιάν, που παρακολουθούσε αυτή τη μελέτη, απεβίωσε λίγο πριν την δημοσίευση. Το λόγο έχει ο κύριος Φεραίρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ για να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Έχετε μπροστά σας τις διαφάνειες, περισσότερο ως οδηγό, δεν υπάρχει κάτι περίπλοκο στις διαφάνειες. So the, the, study was... Λοιπόν, η... σκοπός της μελέτης ε, ήταν να βρούμε πώς αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό τα κράτη-μέλη και τι συνέπειες έχει αυτή η αντιμετώπιση των ε, συμμετοχών και των εσόδων στον τρόπο χειρισμού και διαπραγμάτευσης ε, των ιδιών πόρων. Κάναμε λοιπόν αυτή τη μελέτη και εκ τότε τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Ήταν σημαντική αυτή η μελέτη, παρότι δύσκολη στην ανάγνωση. Ειδικότερα όταν κοιτάμε το τι γίνεται στην κάθε χώρα, διαβάζει κανείς για κάθε χώρα, ε, σε διαφορετικές γλώσσες, διαβάζει τι γίνεται στην κάθε χώρα. Ήμασταν μικρή ομάδα, ήταν δύσκολο το έργο μας. και φυσικά μας έκανε έκπληξη η τρομακτική αταξία που βρήκαμε που διαπιστώσαμε στον τρόπο αντιμετώπισης του προπολογισμού οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αφήνω την έκθεση στον Μάριο Μόντι, στην ε, ομάδα ψηλού επίπεδου για τους ίδιου πόρου. Οπότε τα όσα έχουν από εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μαζί με πολλά άλλα ζητήματα φυσικά. Φαίνεται βαρετή η έκθεση αυτή, αλλά έχει σημαντικέ συνέπειες. Λοιπόν, να περάσω από τα βασικά σημεία της έκθεσης, να μην παραλείψω τώρα την εισαγωγή για τον τρόπο λειτουργίας των ιδιών πόρων, αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα μηνύματα που ε, διακρίνουμε μέσα ε, σε αυτή την έκθεση. Όπως είπα, είναι χαούδης η κατάσταση του σύστημα και θα σας εξηγήσω γιατί αυτό είναι σημαντικό παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ε, της ανάλυσης, ε, της ανάλυσης και των συμμετοχών και των δαπανών. Θα σας παρουσιάσω τις συζητήσεις που κάναμε για τη μεταρρύθμιση της αξινόμησης των πορών και για ποιο λόγο έγινε αυτό, πώς θα μπορούσε μάλλον να γίνει. Επίσης θα ήθελα να συζητήσω λίγο τις επιπτώσεις για τις συζητήσεις για τους ίδιους πόρους. Θα συζητήσουμε λίγο το τι σημαίνει το καθαρό υπόλοιπο όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Θα σας παρουσιάσω κάποιες έννοιες λίγο πιο προχωρημένες ε, ακόμη και από ε, αυτές που εμφανίζονται στην έκθεση γιατί συνεχίζεται η μελέτη αυτών και μετά κάποιες εκθέσεις για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών ε, και πώς αντιμετωπίζονται στον προπολογισμό κάθε χρόνο. Θα ξεκινήσω λοιπόν ε, με την ανομοιογένεια. Τι συμβαίνει. Κοιτάξαμε τους λογαριασμούς του 2014 όλων των κρατών μελών ουσιαστικά. Κοιτάξαμε να δούμε πώς κάνουν τα λογιστικά τους και πώς συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες και πώς καταλογίζουν τις συμμετοχές και τα έσοδα με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, τρεις-τέσσερις χώρες μόνο οι συμμετοχέ στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό δεν ταξινομούνται ω έσοδα που καταλογίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγαίνουν πρώτα στον κρατικό προπολογισμό και μετά καταλογίζονται ω δαπάνη. Ουσιαστικά καμία χώρα δεν εφαρμόζει τον κανόνα του ιδίου πόρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να είναι και η συμβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ουσιαστικά νομικά μπορεί κανείς να πει ότι αν καταλογίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχωρίζεται σαφώ. Ε, από τα εθνικά έσοδα ως έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάτι που γίνεται σε ορισμένες χώρες Τώρα από μια άλλη άποψη, ο τρόπος με τον οποίο τα έσοδα από το υπολογισμό του Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλογίζονται ποικίλει σε σημαντικό βαθμό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να, να παρακολουθήσει κανείς τι γίνεται και δημιουργούνται πολλά προβλήματα διαφάνειας, κόστους και διάφορες δυσκολίες. Ορισμένοι προπολογισμοί, και θα σα δείξω ε, παραδείγματα, σε ορισμένου προπολογισμού δεν υπάρχουν καν έσοδα και συμμετοχέ. Υπάρχει απλά το κόστο διακυβέρνηση τους εθνικού λογαριασμού με κάποιο τρόπο ω ε, επιστροφή γιατί είναι περίεργο γιατί βασίζεται σε υπολογισμό πόρων, δεν είναι επιστροφή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια χρήματα που δεν πηγαίνουν καν στις κυβερνήσεις γιατί πηγαίνουν κατευθείαν στην έρευνα και αυτά. Αλλά υπολογίζεται ως κάτι διαφορετικό. Θα σας δείξω ποιες περιπτώσεις είναι αυτές. Και μετά φυσικά έχουμε και τα ωφέλη των δαπανών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που σπάνια λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να πω ότι από μια όψη αυτό δεν μα εκπλήσει. Το βλέπουμε και στου εθνικού λογαριασμού και στου τοπικού λογαριασμού. Ε, παρατηρούμε πως πριν από εκλογές ε, ή πριν ολοκληρωθεί ένα λογιστικό έτος ε, κάποιοι δρόμοι ξαναστρώνονται σε ορισμένες πόλεις γιατί πρέπει να ξοδευτεί ο προπολογισμό ε, ή κάποιοι τρέχουν δεξιά-αριστερά και ρίχνουν κλήσεις και πρόστιμα για να αυξήσουν τα έσοδα δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά κάποιο όφελος από τη δαπάνη ουσιαστικά οι προπολογισμοί δεν ελέγχουν τη ωφέλη και αυτό είναι ένα πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να πω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και ένα πρόβλημα εθνικό λογαριασμό. Ότι τα ωφέλη και οι δαπάνε δεν λαμβάνονται υπόψη όπω θα γινόταν σε μια επιχείρηση. Ε, εάν οι επιχειρήσει λειτουργούσαν όπω τα δημόσια ταμεία θα κατέρεαν μέσα σε λίγα χρόνια. Αλλά όσον αφορά τι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνουν υπόψη τα κέρδη. Ε, οι προπολογισμοί διάφορων ειδών κέρδη ωφέλη. Ας πάμε στην ταξινόμηση τώρα των ε, ε, συμμετοχών. Οι περισσότερες χώρες τις καταγράφουν ως κρατικές δαπάνες και μόνο στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Βουλγαρία ουσιαστικά καταλογίζονται ορισμένα από τα έσοδα στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό χωρί, χωρίς να θεωρηθούν ε, ε, κρατικές κυβερνητικές δαπάνες, ε, ε κυβερνητικά έσοδα πριν σταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ενδιαφέρον για το ΦΠΑ. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι της Θελωνιακής Ένωσης, τα πράγματα εκεί λειτουργούν κανονικά, αλλά για το ΦΠΑ τα πρα... οι καταστάσεις ποικίλουν. Καταλογίστε με διαφορετικούς τρόπους, γιατί είναι εικονικό ΦΠΑ ουσιαστικά, δεν συνδέεται άμεσα με το πραγματικό ΦΠΑ περιλαμβάνεται στις γραμμές του προπολογισμού με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Οπότε είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αν το θεωρούν δαπάνη. Αλλά πρόκειται για μεταφορά από τον εθνικό προπολογισμό. Οπότε πολύ συχνά θεωρείται δαπάνη παρά ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα έσοδα. Εδώ έχουμε ορισμένε περιπτώσει Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία. Θες, έχουμε εξετάσει όλε αυτέ τι περιπτώσει. Στην περίπτωση του Βελγίου υπάρχει η συμμετοχή που βασίζεται στο ΦΠΑ ως καταλογισμός εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και υπάρχει συμμετοχή βασισμένη στο ΑΕΠ ως ε, δαπάνη. Σε άλλε χώρε ε, καταλογείται σε διαφορετικέ κατηγορίε δαπανών. Οπότε δεν είναι καν οι ίδιες κατηγορίες. Σε άλλες χώρες ε, η συμμετοχή εμφανίζεται ως δαπάνη για διεθνείς οργανισμούς. Σε άλλη χώρα ως γενικές υπηρεσίες. Δεν είναι δηλαδή καν στην ίδια γραμμή του προπολογισμού. Πρέπει να σας πω ότι σε τρελαίνει αυτή η μελέτη, η λεπτομερή όλων των εθνικών λογαριασμών. Και μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο για... δεν εμφανίζεται ούτε καν ως, ε, σωστά ως συμμετοχή. Αυτό που εμφανίζεται είναι μια θεωρητική ε, καθαρή συμμετοχή που εκπίπτει της χοντρικής συμμετοχής ε, όπως αναφέρεται gross contribution και εμφανίζεται ως δημόσια δαπάνη ουσιαστικά στους λογαριασμούς ε, έτσι εμφανίζεται η έκπτωση αυτή το υπόλοιπο εμφανίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς πράγμα που θεωρούμε εμείς εξαιρετικά περίεργο κατάσταση και μετά η Ρουμανία πιθανώ να έχει λάβει συμβουλευτική υποστήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είναι η μόνη χώρα που κάνει το ίδιο πράγμα στα Βαλκάνια. Γιατί άγνωστον. Ε, ίσως να συνεργάζονται. Τώρα πάμε στα έσοδα. Στη Γερμανία τα έσοδα εμφανίζονται μόνο στους ε, εθνικούς λογαριασμούς όταν περνούν από τον εθνικό προπολογισμό. Ουσιαστικά μόνο αυτά τα κομμάτια που πηγαίνουν κατευθείαν στον εθνικό προπολογισμό υπολογίζει, όχι αυτά πάνε στα Λέντερ. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμά τα, όλα τα κονδύλια χωρίς να έχει σημασία ποιος θα παίρνει. Πολύ περίεργο. Ε, η Γερμανία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο δεν θεωρούν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως κάτι, παρότι τα καταγράφουν δεν τα θεωρούν ως έσοδα κρατικά, τα χειρίζονται ξεχωριστά. Δεν ε, περιλαμβάνονται απευθείας στους λογαριασμούς, εμφανίζονται ως ποσό που διακινείται, διαχωρίζουν για άλλη μια φορά εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε πολλές άλλες χώρες ε, αντιθέτως οτιδήποτε λαμβάνεται εμφανίζεται ως εθνικό ε, εισόδημα το οποίο στη συνέχεια δαπανάται. Φυσικά σε διαφορετικές κατηγορίες, με διαφορετικούς τρόπους πρέπει κανείς να δει αναλυτικά σελίδες και σελίδες για να καταλάβει τους λογαριασμούς στην κάθε χώρα. Ε, Συνεπώ για τους ίδιους πόρους τι συμβαίνει. Θα ήταν χρήσιμο, για να μην πω αναγκαίο να υπάρξει κάποια συμφωνία ταξινόμησης των συμμετοχών και των εσόδων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαχωρίζονται από τους εθνικούς λογαριασμούς ώστε τουλάχιστον από γλωσσική άποψη ε, στο πλαίσιο των ιδίων πόρων ε, το ακαθάριστο χώριο προϊόν να θεωρείται ως πόρος αυτό θα βοηθούσε και ανθρώπου σαν εμένα που πρέπει να ελέγξουν του εθνικού λογαριασμού. Θα βοηθούσε ιδιαίτερα για να έχουν μια καθαρή εικόνα. Ο, η χρήση των καθαρών υπολείπων ω δαπανών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διαστρέβλωση. Διότι όταν γίνονται διαπραγματεύσει για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, από τη μία η κάθε χώρα κοιτά τα καθαρά υπόλοιπα Αλλά ξέρετε, αν ολόκληρο το σύστημα των λογαριασμών βασίζεται σε καθαρά υπόλοιπα, πώ να διαπραγματευτεί κανεί με άλλο τρόπο. Δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί τα πράγματα πρέπει να είναι έτσι. Έχουμε δαπάνε και έσοδα, αλλά το να βάζει του λογαριασμού το καθαρό υπόλοιπο ω κρατική δαπάνη δεν έχει νόημα, διότι πολλέ από τι δαπάνε δεν είναι καν τέτοιε. Είναι πιο πολιτική η στάση αυτή παρά λογιστική και κάνει τη μεταρρύθμιση πολύ πιο δύσκολη. Λοιπόν, εδώ λείπει μια λέξη και ζητώ συγγνώμη. Τα πρότυπα για του εθνικού λογαριασμού και τον προπολογισμό τα έχουμε δει και τον υπολογισμό του ακαθάριστου χώρου προϊόντο. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι ομοιόμορφο. Δεν έχουν όλοι πιστεί για την ακρίβεια των υπολογισμών αυτών. Εγώ έβλεπα τι επιπτώσει των ζητημάτων έκπτωση εγώ έχω εξειδικευτεί στον προπολογισμό εδώ και χρόνια και ο καθένα τη εκτό τη υπολογίζει και τα ποσά πρέπει να δοθούν και να επιστραφούν ε, σε επίπεδο ακρίβεια ε, παράξενο. Το ίδιο και με το ΦΠΑ 0, κάτι τη εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο κτλ. Και όταν κοιτάει κανεί τα ποσοστά σφαλμάτων στον υπολογισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο, τρώμε πάρα πολύ χρόνο κάνοντας υπολογισμού που ουσιαστικά ε, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από το ποσοστό σφάλματος. Ελπίζουμε στους επόμενους μήνες να έχουμε μια απάντηση. I was, I was thinking that it, um, Κάτι άλλο που σκεφτόμουν ε, ήταν πρώτα η ταξινόμηση αλλά και ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο προπολογισμό. διότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αιτήσεις διαδικασίες είναι εξαιρετικά περιπλοκή και σκέφτομαι μήπως τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αντιστρέψουν το σύστημα καταλογισμού των εσόδων γιατί ορισμένες φορές τα χρήματα που βάζουν ω συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βασίζεται σε υπολογισμούς πληρωμών ανάληψης υποχρεώσεων και μετά αυτό να έχει ως αποτέλεσμα διενέξεις. Ίσως λοιπόν αυτοί οι καταλογισμοί να μην είναι σωστοί θα μπορούσαν να βασίζονται σε πλήρε υπολογισμού και μετά να υπολογίζονται αντίστροφο, οπότε να αποφεύγονται διενέξεις. Γιατί ξέρετε, ναι, όταν πρέπει να γίνει κάποια πληρωμή, ε, πρέπει να την κάνει το κράτος μάλλον αφού ολοκληρωθεί ένα έργο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για τις μάχες κάθε τρει μήνε για το ίδιο θέμα. Ε, Όπως είπα λοιπόν πρέπει σε κάθε χώρα να διαχωρίζουμε παράλληλα και τους ε, τρόπους αντιμετώπισης των δαπανών και των εσόδων. Ό,τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι είναι εθνικό, εθνικό. Να μην τα αναμειγνύουμε ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Και όπως είπα, η εξάλληψη του καθαρού υπολείπου στο ε, δημοσιονομικά λογιστικά δεν έχει νόημα. Μπορεί αυτό να γίνεται και στους εθνικούς λογαριασμούς ε, και ξέρετε, ο καθένα μπορεί να αρχίσει να τσακώνεται για το ίδιο θέμα, για το καθαρό υπόλοιπα. Εδώ στου εθνικού λογαριασμού δεν λειτουργεί. So what, what is the implication on this? Ποιες είναι οι συνέπειες τώρα για τους ίδιους πόρους, αυτό σκεφτόμουν ορισμένα κομμάτια εδώ, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή γιατί ακόμα ε, τα έχω υπομελέτη. Αλλά είναι ε, σημαντικά στο μέλλον, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα έχουμε κάποιο υπολοιματικό G1, ένα ακαθαριστό εγχώριο προϊόν, ακαθαριστό εγχώριο εισόδημα, συγγνώμη, Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Οπότε είναι σημαντική η σωστή λογιστική και θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, στις μελλοντικές ε, μελέτες ε, για τους πόρους και τις συμμετοχές. Κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό να αμφισβητήσουμε. Δεν μιλάμε πια για ωφέλη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε θέματα εμπορίου, ΑΕΠ ή για συνέπειες. Ο προπολογισμό σήμερα είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι πριν από 30 χρόνια. Όταν κοιτάω του ίδιου πόρου και πώ αντιμετωπίζουν τη χρηματοδότηση στα κρατημέλη και πώ την καταγράφουν, όλα αυτά δεν έχουν νόημα με τη νέα μορφή που αρχίζει να αποκτά ο προπολογισμό. Ε, Επίση έχει πολλά περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση Όλα αυτά, πολλά από αυτά συνδέονται με το σχέδιο Juncker. Ξέρω ότι είναι μόνο για δύο χρόνια, αλλά κοιτάξτε τα ποσά που έχουν κινητοποιηθεί, όχι τι επιπτώσει στο ΑΕΠ και τα ωφέλη του εμπορίου. Τα κράτη-μέλη ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν για τα ωφέλη τα ευρωπαϊκά με αυτόν τον τρόπο, κοιτώντα του ίδιου πόρου. Αλλά ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να τα απασχολεί είναι ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα αυτή εδώ τη περίοδου συμπεριλαμβάνουμε το, συμπεριλαμβάνουμε ότι ε, υπάρχουν και οι διασφαλίσει ε, οι δημοσιονομικέ του σχεδίου Juncker. Μιλάμε για εκατοντάδε δισεκατομμύρια ευρώ παράλληλα ω επενδύσει, ένα σχέδιο το οποίο πιθανότατα θα δημιουργήσει εισοδήματα, θα ε, φέρει αποτελέσματα. Πρόκειται λοιπόν για επενδύσει και τέτοιε ροές, τέτοιε χρηματικές ροέ εντό αυτών των μέσων ε, δεν μπορούν να έχουν διαφορετικά καθαρά υπόλοιπα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ουσιαστικά, ποιοι επωφελούνται από το σχέδιο Juncker. Έχουμε δει διάφορα. Έχουμε δει το φυσικό αέριο στην Ισπανία, κάποια άλλα στι βόρειε χώρε. Μιλάμε για κίνηση εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων που επηρεάζονται από τον ευρωπαϊκό υπολογισμό και εμεί αντί να δω, βλέπουμε αυτά τα χρήματα, καθόμαστε και κοιτάμε τα καθαρά υπόλοιπα. μπορεί να μιλάμε και για 700 δισεκατομμύρια ξέρετε, που θα κινητοποιηθούν στο, στο, σε όλους τους τομείς για αυτό το διάστημα για όλα τα μέσα. Μιλάμε ουσιαστικά ουσιαστικά αναφερόμαστε σε τέτοια ποσά όπως ε, αντιμετωπίζουμε και τον υπολογισμό των καθαρών υπολείπων. είναι σαν να παίρνουμε ένα ευρώ από τον ε, προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίρνουμε και ένα ευρώ από τον εθνικό προπολογισμό και να λέμε ανακινητοποιήσαμε ε, χρήματα, υπολογίζουμε ε, τα ωφέλη. Δεν, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό πλέον. Δεν έχει νόημα. Και στο τέλος έκθεση, όπω έχω πει, αναφέρω την ετήσια δημοσιονομική διαδικασία είναι καλύτερο να υπάρχουν καλύτερε λογιστικέ διαδικασίε ώστε να απαλληλθούν οι εντάσει. Τα τελευταία χρόνια οι εφημερίδε αναφέρονται στο ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτό ελέγχου και οι ηγέτε και ευρωπαϊκών χωρών λένε το ίδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι για λόγους έρευνας και για να διατηρήσουν και ερευνητές όπως εγώ ε, ε, τη λογική τους και να μην τρελαθούν. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο να ε, καταρτίζουμε τους λογαριασμούς. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή, η οποία δείχνει πράγματι ότι υπάρχει ανομοιογένεια. Πρώτα απ' όλα στο πώς υποβάλλονται οι δημόσιοι λογαριασμοί από τα διάφορα κράτη-μέλη και συνεχεία σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή των συνεισφορών των κατάμελων ε, ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, στους εθνικούς λογαριασμούς. Είναι ε, κάπως ε, μοναδική αυτή η κατάσταση, δηλαδή ότι ναι τα κράτη μεν συμμετέχουν, αλλά δεν έχουν φροντίσει να παρουσιάσουν τον ίδιο τρόπο τις συνεισφορές. Θα επανέλθουμε βέβαια. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. ίσως αναλάβει τις ευθύνες της Eurostat. Βέβαια δεν έχει και πολλά μέσα στη διάθεσή της. Στα μακροοικονομικά τα πάνε πολύ καλά, αλλά για να επαληθεύσουν ε, την ειλικρίνεια των ε, λογαριασμών, των εθνικών λογαριασμών, έχουν πολύ λίγο προσωπικό. Είναι ένα είδος γενικής διεύθυνσης ε, ελεγκτών της Ένωσης. Έχουν πάρει τρεις θέσεις παραπάνω αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ περισσότερο τα πράγματα. Γιατί οι λογαριασμοί δεν παρουσιάζονται με τρόπο εύληπτο για τους ε, πολίτες μας. Έρχομαι στον κύριο και το μόνιμο εισηγητή που δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Τότε να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπρέ που είναι παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και με προσήλωση ενίοτε το κείμενο γιατί κάποιες σελίδες ε, που αναφέρονται στην κατάσταση των κρατών μελών ε, μου δημιούργησαν κάποια ενόχληση, ας πούμε κάποια προβλήματα. Έχω τρία ερωτήματα. Το πρώτο. Συμφωνώ με τους συντάκτες της έκθεσης που υποστηρίζουν ότι πρέπει να εναρμονιστεί ο καταλυσμός ε, των εισφορών των κρατών μελών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ονοματολογίας. Ε, ένα θέμα που με έχει απασχολήσει γιατί έχω εργαστεί πολύ για τον προπολογισμό στη χώρα μου και όταν καταρτίζουμε στο Βέλγιο, να σας δώσω το παράδειγμα της χώρας με τον προπολογισμό, προβλέπουμε έσοδα και ένα μέρος αυτών των εσόδων τροφοδοτεί την συμμετοχή, την συνεισφορά του Βελγίου στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αφελώ ή ε, ανοήτως αν θέλετε, είναι δαπάνη για το Βέλγιο αυτό. Ε, αυτή η συνεισφορά. Θέλω να εξηγήσετε λοιπόν με ποια συλλογιστική εσεί, αν κατάλαβα καλά, κάνετε μια διαφορετική πρόταση και τι όφελος θα μπορούσε να συνεπάγεται αυτός ο διαφορετικός καταλογισμός και σας τα λέω επειδή έχω εμπειρία. Έχουμε λοιπόν έσοδα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά με αυτά τα έσοδα κάνουμε κάποια εμβάσματα, πληρωμές, ε, μεταφορές πιστώσεων κτλ. Δεύτερο, αν κατάλαβα καλά, αυτά που είπατε για τα έσοδα της Ένωσης ε, που πηγαίνουν από τον προπολογισμό του εθνικού στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Δεν κατάλαβα καλά. Προτείνεται εναρμόνιση. Όχι, από ό,τι κατάλαβα. Αφήνεται δηλαδή πιο πολλά περιθώρια, μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη χρήση της ονοματολογίας και τον καταλογισμό. Γιατί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ε, γίνεται διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τα έσοδα. Τώρα, ήδη οι Πάλι δεν ξέρω να κατάλαβα καλά. Αν συνοψίζω σωστά την πρότασή σας, μπορούμε να έχουμε ιδίους πόρους. Εσείς έχετε μία προτίμηση για το ΦΠΑ, είναι προφανές. Όμως λέτε σε κάθε περίπτωση ότι θα πρέπει να υπάρχει παραπέρα και ίσως σε ένα πρώτο χρόνο φαίνεται να είστε υπέρμαχοι του να έχουμε ένα σύστημα που ήδη οι πόροι θα είναι εισφορές των κρατών. Λάθος, κατάλαβα, έτσι μου φάνηκε ότι είπατε. Δηλαδή σε ένα πρώτο χρόνο, αν έχουμε εναρμόνιση ε, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δημοσιο... Ε, ονοματολογίας για το καταλογισμό των εισφορών των ε, κρατών μελών στον προπολογισμό της Ένωσης, θα μπορούσαμε τις εισφορές των κρατών μελών με βάση το καθάριστο εγχώριο εισόδημα, να τις θεωρήσουμε ως ίδιο πόρο. Και σε μια δεύτερη φάση, αν κατάλαβα πάλι καλά, και ακόμη δυσκολεύομαι να κατανοήσω τη συλλογιστική σα, όταν θα έχουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων που θα βασίζεται στο ΦΠΑ, θα πρέπει, ε, από ό,τι φαίνεται, να διατηρήσουμε μια θέση για τις ε, συμμετοχές των χωρών, για τις ε, εθνικές συνεισφορές. στο πλαίσιο μιας οικονομικής χρήσης. Χρειάζονται περισσότεροι οικονομικοί πόροι και δεν καλύπτεται αυτό από το ΦΠΑ. Πρέπει κάπου να αναζητήσουμε τους επιπλέον αυτούς πόρους, γιατί δεν μπορούμε τους συντελεστές του ΦΠΑ εν μέσω της οικονομικής αυτής χρήσης να τους τροποποιήσουμε. Αυτή είναι πράγματι η συλλογιστική σας πίσω από αυτό που εγώ τουλάχιστον ερμηνεύω ως πρότασή σας αυτά σε αυτή την φάση κύριε Πρόεδρε. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου και οι ερωτήσεις μου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε στον εισηγητή μας. Ναι, ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα αγγλικά ε, λόγω της ορολογίας. Λοιπόν, όσον φορά την αναρμόνιση και τον τρόπο συμμετοχής. Η Γαλλία και άλλες χώρες είναι εκείνες που καταλογίζουν τη χρηματοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας το ίδιο πρόβλημα. Ταξινομούν τα χρήματα την ώρα που τα εισπράττουν και τα καταγράφουν ως ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά το θέμα είναι να υπάρχει μια σαφής γραμμή προϋπολογισμού αντί να υπάρχει μια γραμμή ε, εσόδων και μετά οι συμμετοχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε κάθε χώρα. Οπότε είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανεί τι γίνεται. Δεν χρησιμοποιούν όλε οι χώρε την ίδια γραμμή του προπολογισμού για να ε, καταλογίσουν τα, τα ε, συμμετοχέ αυτέ. Δηλαδή είναι ουσιαστικά σκοπό μεγαλύτερη διαφάνεια, να ξεχωρίσουν ε, από τι υπόλοιπε δαπάνε τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κατάλαβα καλά, για να μην υπάρχει παρανόηση, θέλετε μία συγκεκριμένη γραμμή στον προπολογισμό που να σημαίνει το ίδιο πράγμα στους προπολογισμού όλων των κρατών μελών. Αυτό ζητάτε, μάλιστα. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό που συμβαίνει σε μια χώρα όπως η Γαλλία, στα σχέδια προπολογισμού, θέλετε να εμφανίζεται το σύνολο των ε, ε, δημοσιονομικών πόρων και πριν οριστεί το ποσό των εσόδων που θα διαθέσει το κράτος αφαιρούμε την συμμετοχή που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα εμφανίζεται ως δαπάνη, θα εμφανίζεται ως ε, μεταφορά ε, δημοσιονομικών εσόδων προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκεί καθορίζουμε το ποσό το οποίο θα διαθέσει, θα έχει στη διάθεσή του το κράτος μέλος αφού εισπράξει τους φόρους εκ των οποίων ένα κλάσμα πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσθέσω και κάτι ακόμη. Στη Γαλλία χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία για τον καταλογισμό και στον περιφερειακό προπολογισμό. Δηλαδή και σε εθνικό επίπεδο θα βοηθούσε να υπάρχει ένα σύστημα για να γίνεται πιο σαφές. Όταν ο φόρος ο πόρος είναι σχεδιασμένος για να χρηματοδοτήσει το περιφερειακό επίπεδο. Να φαίνεται αυτό. Για να έχουμε ευλήπτους και διαφανείς εθνικούς λογαριασμούς. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Είπατε επίσης πώς ε, χειριζόμαστε τις δαπάνες τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε να υπάρξει εν μέρη μια εναρμόνιση, αλλά τα πράγματα εκεί είναι πιο πολύπλοκα, γιατί δεν παίρνουν όλα τα κράτη-μέλη χρήματα για τους ίδιους σκοπούς. Θα μπορούσε ίσως να υπάρξει κάποια διευκόλυνση, αλλά νομίζω ότι εμείς επειδή εστιάζουμε τώρα στις συνεισφορές και γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί επηρεάζουν πραγματικά ε, τις διαπραγματεύσεις για τους ε, πόρους. Αρχικά η μελέτη είχε ως αντικείμενο όχι τόσο να δει ε, πώς ε, επηρεάζονται αυτές οι συζητήσεις, ο πρόεδρος Αρτουή, υπάρχει ένα πρόβλημα για το κλείσιμο ε, των λογαριασμών, γιατί δεν είναι η ίδια ημερομηνία σε όλες τις χώρες. Έχετε δίκιο, ο κύριος Φερέρ. Για το ΦΠΑ. Έχουμε συμπεριλάβει το ΦΠΑ στη μελέτη μας. Μας ζητήθηκε να πούμε ε, τις απόψεις μας. Είναι μια επιλογή. Ο ίδιος σπόρος αλλά ίσως θα το δούμε πιο αναλυτικά στην επόμενη μελέτη μας, γιατί εδώ δεν το αντιμετωπίσαμε σε βάθος. Είναι χρήσιμος ο ΦΠΑ πάντως, όμως ό,τι αφορά το καθάριστο εισόδημα, δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί και τόσο εύκολα μπορεί πράγματι να είναι χρήσιμο όταν πρέπει να αλλάξουν προτεραιότητες. Ένα πρόβλημα με τον προπολογισμό είναι ότι μας επηρεάζουν πολλά στον κόσμο και θα πρέπει τον προπολογισμό να τον μελετούμε σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Άρα ο πόρος αυτός, το καθαρίζω εθνικό μπορεί να είναι ένα χρήσιμο ε, εργαλείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και επίσης μπορεί να είναι απαραίτητος ο πόρος αυτός για την ε, εξάλληψη κάποιων ε, μεγάλων διαφορών ε, που μπορεί να έχουν κάποιοι σε, ως προς τις απόψεις για διάφορους ιδίους πόρους. Επίσης, ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει πολλές επιπλέον αναλήψεις υποχρεώσεων δεσμεύσεις, οι οποίες δεν είναι καταγεγραμμένες. Αυτό σημαίνει ότι εγγυάται αυτός ο προπολογισμό με περιθώριο ε, ένα ισοζύγιο πληρωμών ή έχουμε ε, άλλα κονδύλια για την Ελλάδα και για, άλλους, για άλλες χώρες. Αν υπάρξει πτώχευση, χρεοκοπία μιας χώρας, θα πρέπει να καταβληθούν κάποια χρήματα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι πάντα θα υπάρχει αυτός ο πόρος, ο πρόεδρος. Ναι, είναι εκτός, ε, αν θέλετε, ισολογισμού αυτές τι δαπάνε. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε πώς θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό ε, αυτές τις ενισφορές εκτός ισολογισμού. Ε, κύριε Ραποβησηγητά. μετά από αυτά, νομίζω ότι υπάρχει ένα διαφορετικός αντίκτυπος για αυτά που λέγαμε, δηλαδή μηχανισμός εγγύσεων εντός κρατών ακόμη και εκτός λογισμού. Πώς θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό, γιατί εδώ βλέπω ε, να υπάρχει μια διαφορετική λογική. Υπάρχουν πόροι, υπάρχουν έσοδα και δαπάνες τέλο πάντων. Οι εγγυήσεις μπορεί να γίνουν ε, δαπάνες. Δεν μπορούν αυτά να μπουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί μόνο οι χώρες της Ευρωζώνης ε, συμμετέχουν. Ναι, υπάρχει προπολογισμός τη Ευρωζώνης λέει ο κύριος Αρτουή. Θα ήταν μια ιδέα. Ε, ναι, θα ήταν καλό, λέει ο κύριος Είναι που το, το συζητάμε μαζί με διάφορα άλλα μελλοντικά ζητήματα. Το πώς θα χειριστούμε τα ζητήματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Το ESFM εγγυάται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, το ισοζύγιο πληρωμών και έχουμε και την ελληνική περίπτωση. Γι' αυτό είχαμε και μια εξαίρεση για το ε, Βρετανία. Έλαβαν ένα δάνειο 7,5 δις που εγγυάται από το περιθώριο του προπολογισμού μεταξύ των πληρωμών και του ανωτοτού όριου. Αν πάει τι ή άσχημα, το Ηνωμένο Βασίλειο λέει δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Ε, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα υπάρχει ένας μηχανισμός για το πώς θα καλυφθεί μια αδυναμία πληρωμών. Δηλαδή, κανονικά λέμε ότι μια χώρα που έχει αδυναμία πληρωμών πρέπει αυτή να την καλύψει. Και τα απαντάει το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω, λέει το Κοινοβούλιο το Βρετανικό, ότι συγγνώμη δεν υπάρχει μηχανισμός αν μια χώρα ε, κηρύξει στάση πληρωμών. Αν, ακόμη και δεν είναι Ευρωζώνη, ας πούμε ότι είναι η Ουγγαρία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληρώσει αλλά θα λάβει έκπτωση διότι δεν διαφοροποιούνται οι δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ε, προβλήματα όσον αφορά αυτό το περιθώριο τα οποία όμως θα επιληθούν ε, θα συνεχίζουμε και τα μελετάμε τώρα με ρωτάτε αν θέλουμε να τα διατηρήσουμε όλα, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, αν θέλουμε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα είναι καλός πόρος, εξαρτάται. Εμείς το σκεφτόμαστε εντατικά αυτή τη στιγμή. Έχει κάποια καλά πράγματα το καθαρό στο εθνικό εισόδημα. Όταν ε, φτιάχνει κάποιος, ξέρετε, ε, ε ιδίους πόρους ε, για το μέλλον, μην νομίζετε ότι ο κόσμος θα είναι ευκολότερος. Θα είναι διαφορετικός, αλλά θα εξακολουθούν να υπάρχουν διενέξεις για τα ποσοστά, για όλα αυτά. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι το καθαρό στο εθνικό εισόδημα έχει κάποια πλέον εκτήματα γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος και για την αντιμετώπιση έκτακτων προσθετικών ενώ άλλοι διπόροι είναι καλοί για άλλα ζητήματα. Κάτι λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πόρο ο οποίο να ευθυγρομίζεται με κάποιο συγκεκριμένο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, υπάρχει δηλαδή αυτή η δημοσιονομική επιρροή ω εξουσία των κρατών μελών. Δηλαδή, ο πόρο να κάνει κάτι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ευθυγραμμίζεται με ένα στόχο, αλλά μετά να νομίζουμε ότι ο πόρο θα υπάρχει εκεί χωρί οι χώρε να ξέρουν τι πληρώνουν. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν θέλω να κριτικάρω δηλαδή ω κακό το ακαθάριστο εθνικό ζώδημα. Από τεχνική άψη. δεν είναι άσχημο. Κύριε Ντεπρέ. Πανέρχομαι στην ερώτησή μου. Ας υποθέσουμε ότι αύριο, εκτός από του φυστάμενου ίδιου πόρου, αποφασίσουμε για έναν νέο ίδιο πόρο, που υποθέτουμε ότι είναι ασχετικό ποσοστό του ΦΠΑ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό ΦΠΑ ορίζεται στην αρχή του οικονομικού έτους, της υποθέσουμε ότι ε, στο πλαίσιο εκείνη τη οικονομική χρήση έχουμε μια μεγάλη καταστροφή και αυτό επιβάλλει την κινητοποίηση περαιτέρω κονδυλίων. Ο πιο απλό πόρο αντί να τροποποιηθούν συντελεστέ του ΦΠΑ και να περάσουμε σε απόλυτη διαδικασία και τι επιπτώσει που θα έχει αυτή, ο πιο απλό τρόπο θα ήταν, επαναλαμβάνω, να ζητηθεί μια πρόσθετη συνεισφορά ε, σε συνάρτηση πάντα με το ε, εισόδημα, το εθνικό ακαθάριστο εισόδημα. Άρα λέω, με τον έναν τον άλλο τρόπο θα είναι ένα έσχατο καταφύγιο, μια έσχατη λύση η κινητοποίηση αυτού του πόρου. Απάντηση. Άλλες λύσεις δεν έχω. Ε. Πρόεδρος, η πτυχή, το σκέλος ε, έσοδα σας διαφεύγει. Υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ των μελών που συμφωνούν ε, μετά από κάποιες διαπραγματεύσεις και έχουν μια μικρή επιστροφή στο ΦΠΑ και τα λοιπά. Γίνεται ε, ένα παζάρεμα, αν θέλετε, μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς δεν έχουμε ιδέα για όλα αυτά στο Κοινοβούλιο. Τώρα τι γίνεται με το ΦΠΑ, με το καθάριστο εθνικό εισόδημα. Το θέμα είναι ε, πώς θα πληρώσει ο Γιώργος και όχι τόσο ο Κώστας ή ο Χρήστος. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ λέω τώρα, είτε είναι ο ΦΠΑ, είτε είναι ε, κάποιοι φόροι πάνω στα έσοδα ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι αφαιρούμε από τα φορολογικά έσοδα ε, της κάθε χώρας ένα ποσοστό για τη συμμετοχή της στον εθνικό προπολογισμό. Αλλά είναι πραγματικά ε, πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις και ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο κάποια στιγμή θα πρέπει να συμμορφωθεί σε ένα γενικότερο κανόν. Ο κύριος Εντονανό πάρα πολύ σύντομα και ο κύριος Μάνκα. Ναι κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την έκθεση. Χαίρομαι που ήρθα σήμερα το πρωί μου. Μου κάνει μεγάλη έκπληξη τα όσα υπόθηκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να έχουμε φτάσει εκεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την οργάνωση των εσόδων των ε, κρατών ε, είναι ανήκουστο το να μην έχουμε βρει πιο διαφανείς τρόπους για τη συμμετοχή των κρατών μέλων διότι ξέρετε αυτό επηρεάζει πολλούς τομείς ένα από τα ερωτήματα που έχω είναι αυτό επηρεάζει Αυτό ο υπολογισμό των συμμετοχών των κρατών επηρεάζει αυτό το γνωστό το 3% της σύγκλησης ε, διότι όταν συζητάμε για την εσωτερήκευση των δαπανών ε, θα πρέπει, των εσόδων, συγγνώμη, αυτό θα πρέπει να έχει κάποια επίπτωση. Και με τα πολύ ειλικρινά υπάρχει και όλο το ζήτημα των απατών, της απάτης που τελικά υπάρχει η απάτη με το ΦΠΑ, η απάτη με το καθάριστο εθνικό εισόδημα και όλο αυτό μου φέρνει δάκρυα. Οπότε πιστεύω είναι επίγον να βρούμε σήμερα τρόπους χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο διαφανείς. Οπότε εγώ περιμένω με μετέρα ε, η όβια υπομονή να δω τις νέες σας προτάσεις, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε νέους ε, πιο ισότιμους ε, τρόπους δημιουργίας εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε ποιος πληρώνει τι, οπότε υπό το πρίσμα της διαφάνειας θα ζητώ όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τελανό που εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Ο κύριος Ροκά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σίγουρα χρειάζεται κάποια ε, εναρμόνιση. Κάποιες χώρες αποσιάζουν από αυτή την έκθεση. Τα constat ou une interrogation, Λοιπόν, η χώρα μου δεν έχει συμπεριληφθεί. Τι σημαίνει αυτό ότι οι χώρες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση είναι εντάξει. Γιατί ξέρετε, στη χώρα μου υπάρχουν ορισμένε πόλεις και κάποιοι δήμοι που είναι καθαροί αποδέκτες μόνο εισπράττουν και κάνουν τα λογιστικά τους ακριβώς όπως και οι επιχειρήσεις. Τώρα αναφέρθηκε το ΦΠΑ και θα ήθελα να αποδείξει. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών. Ε, στην μια χώρα 10, στην άλλη 25%. Οπότε σίγουρα χρειάζεται και εναρμόνιση εδώ πέρα. Διότι αυτοί που πληρώνουν 25% ε, στο εθνικό σύστημα δίνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνονται σε άλλες χώρε όπου το ΦΠΑ είναι ας πούμε μόνο 10%. Τώρα όσον αφορά την έκθεση για τους ίδιους πόρους το ΦΠΑ αναφέρεται ως ε, ε, βάση κλειδί των εσόδων και φυσικά το ΦΠΑ είναι και χαρακτηριστήκε από μεγάλη φοροαποφυγή όπως γνωρίζουμε οπότε θα προτείνουμε το ΦΠΑ να πληρώνεται από αυτούς που βρίσκονται στο τέρμα της οικονομικής αλυσίδας έτσι ώστε να αποφεύγεται ε, μεγάλο ποσοστό αυτών των απατών Ξέρετε το ΦΠΑ περιλαμβάνει πολλές γκρίζες περιοχές και πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να πληρώνουν το ΦΠΑ αυτοί που βρίσκονται στο τέλος της αλυσίδας. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάνκα για την ιδέα αυτή μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ. Να έχουμε ένα ομοσπονδιακό ΦΠΑ. Ο κύριος Τάραντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και όλοι και εγώ εκτιμώ πολύ την προσέγγιση της έκθεσης αυτής. Και είναι απόλυτα λογικό το ότι προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Θα ήθελα όμως να πάω και λίγο παραπέρα, γιατί μου φαίνεται πως, μου φαίνεται πως είμαστε σε μή, όπως οι λογιστές στους Monty Python. Εστιάζουμε στους ιδίους πόρους, στο ευρωπαϊκό εισόδημα και τα κράτη-μέλη συνεχίζουν αυτή την πρακτική που είναι δυσνόητη από εμάς. Από εμάς και όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους ψηφοφόρους μας στην Ευρώπη. Προσωπικά θεωρώ πως ένας άμεσος ευρωπαϊκός φόρος, ε, πέρα από το ΦΠΑ, το οποίο είναι και αυτό μια καλή προσέγγιση, αλλά όταν όλοι οι πολίτες πληρώνουν, παραδείγματο χάρη, ένα ευρώ το χρόνο, είναι ένα μικροσκοπικό ποσό σε σχέση με τους φόρους που πληρώνουμε στα κράτη-μέλη. Θα έχουμε αμέσως 450 εκατομμύρια. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρώπη, γιατί με αυτά τα χρήματα μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όταν λοιπόν οι πολίτες συμμετέχουν, έστω και λίγο, είναι πολύ ωφέλιμο είναι κάτι που δεν το αισθανόμαστε τώρα, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα έσοδα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Θεωρώ προσωπικά πως ε, πρέπει να αρχίσουμε με μικρά βήματα. Καταρχάς πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι χρήματα έχουμε εξοδέψει σε αυτές τις ε, υψηλόβαθμες ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του Μάριο Μόντι τα τελευταία χρόνια και τι έχουμε πάρει από αυτά, με αυτά τα χρήματα που έχουμε πληρώσει. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε κύριε Τερόν. Θα δεχτώ ο μιλητής, ο πρόεδρος της αυτός. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Ινιασφαιρέα ε, για αυτή την παρουσίαση και χαίρομαι που τα δημοσιονομικά θέματα μπορούν να δημιουργήσουν ε, συναισθήματα. Μιλάμε για αυτά τα θέματα πάντα από τεχνική άποψη και πρέπει να βγούμε από αυτό το πλαίσιο. Σήμερα είναι αναγκαίο να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να παρουσιάζουν τους δημόσιους λογαριασμούς τους με τρόπο ομοιογενή και ευανάγνωστο, κατανοητό Δεν ξέρω αν πρέπει να διαχωρίζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια από του εθνικού προπολογισμού ή να εγγράφονται ω εθνικέ δαπάνε, αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσουμε επί μια μεθόδου. Αυτό ο διαλόγο μεταξύ των κρατών μελών έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Μιλάμε για αυτό το 3% για τα δημοσιονομικά θέματα, για το πόσο σπουδαία είναι όλα αυτά. Δεν πρέπει η Επιτροπή μα κύριε Σιγητά, να εκφράσει κάποια είδους ευχή υπό τη μορφή κάποιου ψηφίσματος όπως η, τα Υπουργεία Οικονομικών, ε, τα ταμεία του κάθε κράτου μέλους να καθίσουν να δουλέψουν για να εναρμονίσουν τους δημόσιους λογαριασμούς και για να συμφωνήσουμε μία ίδια μέθοδο παρουσίασης ε, της συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και το πώ αυτό θα εμφανίζεται ίδια παρουσία στου εθνικού Προπολογισμού Δεν ξέρω, μπορείτε να λάβετε εσεί κάποια πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συζήτηση, να το συζητήσουμε καθαρά, να ζητήσουμε από την Eurostat να έρθει και να μα πει τι μέσα υπάρχουν, τι ομάδε εργασία μπορούν να οργανωθούν, ώστε να πετύχουμε ε, κανόνες ε, δημοσίων ε, λογιστικών ίδιους. Αλλιώς τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Το ελεγκτικό συνέδριο που ελέγχει την ορθότητα των εθνικών λογαριασμών θα πρέπει έτσι να μπορεί να εξετάσει τα πράγματα με ομοιόμορφο τρόπο και να καταλαβαίνει ποια είναι τα αποτελέσματα και πόσο αποδοτικά είναι τα κράτη-μέλη. Είναι αναγκαίο λοιπόν πιστεύω να εκφράσουμε ε, με σοβαρότητα και με επιμονή ε, αυτή την αναγκαιότητα. Αλλιώς όσο και να καλοπίζουμε τα δημοσιονομικά δεν θα καλύψουμε την ανηλικρίνεια των λογαριασμών. δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο αντί να βάζουμε τα πράγματα συνέχεια κατά το χαλί στην τουλάπα. Να γίνει κάτι. Εσείς μαζί με τον κύριο Λεβαντόφσκι δεν μπορείτε να λάβετε την ευθύνη να ε, κάνετε μια παρέμβαση. Ας ακούσουμε και τις απαντήσεις τους ε, διαφορούς ομιλητές και μετά να κλείσουμε. Ναι, λοιπόν ευχαριστώ θα χαρείτε μαθαίνοντας ότι με προσέγγισε όχι θεσμός αλλά διάφοροι απελπισμένοι άνθρωποι δεν θα κατονομάσω κανέναν τώρα προετοιμάζουμε μια ειδική ομάδα υψηλού επίπεδου για τους δημόσιους λογαριασμούς με εξειδικευμένο προσωπικό από ολόκληρο τον κόσμο για να συζητήσουμε το ζήτημα των λογαριασμών. Συζη δείτε στην Ευρώπη το ΕΨΑ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δημοσίων Λογαριασμών, αλλά τα πράγματα δεν κινούνται. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα στην κάθε χώρα και ακόμα και ο τρόπο καταχώρηση δεν δείχνει καθαρά τι εισόδου και τι δαπάνε. Υπάρχει και μια χώρα που έχει διπλού λογαριασμού, μεσονικέ καταστάσει. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα όταν μιλάμε για τέτοια και μετά πρέπει να καθόμαστε να σώζουμε χώρε και τέτοια. Δηλαδή Αυτά, είναι αυτά είναι που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον, ε, να το ξέρετε. Τώρα, ε, πολύ γρήγορα για το ΦΠΑ. Όπως ξέρετε το ΦΠΑ ε, είναι μία ποσοστιαία μονάδα του πραγματικού ΦΠΑ οπότε τα πράγματα υπάρχουν, είναι διαφανή. Το ζήτημα της γκρίζας ζώνης είναι ζήτημα. Σε κάποιες χώρες το ποσοστό σφάλματος είναι 2% και σε άλλες είναι γύρω στο 20% το ποσοστό σφάλματος αυτό το πόσο χάνεται ουσιαστικά είναι σοβαρό το ζήτημα τώρα όσον αφορά το 3% και κατά πόσο αυτό επηρεάζει το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Αλλά πράγματι ε, στα συστήματα λογαριασμών κανονικά οι δαπάνες και τα έσοδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι δαπάνες ουσιαστικά συνυπολογίζονται με τα ελλείμματα του προϋπολογισμού ε, υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις αλλά υποθέτω ότι επειδή ο προϋπολογισμός ε, έχει άλλες πτυχές εκτός από το πραγματικά 3% υπάρχει κάποια επίπτωση αλλά δεν την έχουμε υπολογίσει ε, χρειάζεται ειδικού υπολογισμού οπότε εκεί είναι ένα ζήτημα And, Direct taxes. Uh, Τώρα για τους άμεσους φόρους, ε, ξέρετε, είχαμε σκεφτεί κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και με διαφάνεια μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής. Απλά μπαίνει στο φόρο του κάθε ατόμου ότι, ξέρετε, τόσο ποσοστό είναι συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και να πείστε αυτό που δεν το έχουμε κάνει. Αλλά, ξέρετε, τα περισσότερα κράτη-μέλη όμως δεν το θέλουν. Δεν τους αρέσει ανέκαθεν υπήρχαν τέτοιες επιλογές διαφανείς ε, για να αντιμετωπίσουμε τους σπόρους ε, αρκεί να έχουμε το κατάλληλο κουτάκι ε, αλλά πραγματικά κανείς δεν προσπαθεί να έχουμε ομοιογένεια όλοι προσπαθούν να έχουμε ετερογένεια τώρα η ισορροπία μεταξύ ε, ε κόστους και εσόδων ελπίζω τα χρήματα να έχουν δαπανηθεί σωστά La conclusion pour Monsieur Depré. Αφήνω τον κύριο Ντεπρέ να διατυπώσει τα συμπεράσματά του. Τα σημείωσα όλα κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και τη δική σας υπόδειξη και θα δώσω συνέχεια. Κατά τα λοιπά, απλά κλείνω έτσι, μια ευθυμινότητα αυτήν την παρουσίαση. Να σα υπενθυμίσω, λέει πρόεδρο, ότι ο κύριος Μόντι δουλεύει, εργάζεται. Ε, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά η ομάδα του εργάζεται. Και υπάρχουν σε αυτήν την ομάδα Μόντι και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα έρθουν εδώ. Και μάλιστα στις 19 Νοεμβρίου. Θα είναι μια μεγάλη στιγμή. Πολλά υποσχόμενη. Και ο κύριος Ντενανό ίσω κατευνάσει με αυτόν τον τρόπο και τι ανησυχίε του. Είδατε τι ωραία. Λοιπόν, Κυρίες και κύριοι, αυτά, αλλά δεν είναι παρά η αρχή. Είμαστε στην αρχή ενός μιας μακράς πορείας. Διότι αν εμείς οι ίδιοι δεν ασχοληθούμε με την τυποποίηση των ε, λογαριασμών, θα το κάνουν άλλοι. Σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τα σχετικά πρότυπα, το EFRS είδατε τι έγινε εκεί. Το θέμα είναι να έχουμε σαφείς λογιστικές αρχές οι οποίες θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη με την παρουσίαση των ε, δημόσιων λογαριασμών διότι δεν έχουμε την εντολή ε, ουσιαστικά να λογοδοτούμε για τις δράσεις μας στα κράτη-μέλη. Τώρα, ας περάσουμε στην δόκτωρα Φιώνα Μπέβεριτς και στον δόκτωρα Φιρά Τσενγκίζ που θα μας παρουσιάσουν τους καρπούς ε, των εργασιών τους. Ε, πρόκειται δηλαδή για την παρουσίαση της μελέτης με θέμα ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Η έκθεση, η μελέτη ανατέθηκε από την Επιτροπή Γυναικών. Θα μελετηθεί, μελετήθηκε τέλος πάντων ο της Ένωσης με βάση έξι τομείς, πάντως όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Κάτι που δεν βλέπουμε να είναι πάντοτε δεδομένη. Θέλουμε καλύτερη χρήση των δικτών που σχετίζονται με τα φύλλα και πιο συστηματική ε, συλλογή δεδομένων κατανεμένων ανά Έχουμε τη μελέτη στα αγγλικά, γαλλικά και στα γερμανικά εδώ στην αίθουσα. Η κοινοπραξία Blom Γιορενσάνζη κάπως έτσι ανέλαβε να καταρτήσει αυτή τη μελέτη. School of Law and Social Justice Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ ήταν ένας από τους συμμετέχοντες. Η Dr. Beveridge που είναι στο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών ε, στο Λίβερπουλ ειδικεύεται τα κοινωνικά ζητήματα και δει στην ισότητα των φίλων και έχει δημοσιεύσει πολλαπλά άρθρα. Ο κύριος Σεντζής είναι μέλος Πανεπιστήμιου του Λίβερπουλ και αυτός και αναφέρει σε διάφορους τομείς, ε, τα, την πολυεπίπεδα δίκτυα. Θα σας δώσω το λόγο η Πατρίσια Σουλίν παρακολουθεί το Gender Mainstreaming Network και θα λάβει το λόγο μετά τους προσκεκλημένους ή τις προσκεκλημένες, δεν έχουμε καταλάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που μου έδωσε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φίλων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας ήταν να εξετάσουμε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η συνεκτίμηση της ισότητας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσουμε μια μεθοδολογία για να δείξουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός λειτουργεί προς όφελος Τη ε, πρόθεση τη ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, έρευ, μελέτη αυτή διεξήχθη ανάμεσα στον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2015 και ω επιτοπλίστων ήταν μια δευτερογενή στατιστική ανάλυση με συνεντεύξεις με διάφορου ε, ενδιαφερόμενους και ε, υπαλλήλου Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια μεθοδολογία που να μα αποφέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη μου χαρά σήμερα μπορώ να σα παρουσιάσω τα αποτελέσματα τη μελέτη μα. Το ερώτημα λοιπόν του γιατί χρειάζεται συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό. Γιατί χρειάζεται και πώς μπορεί να μας ωφελήσει. Η συνεκτίμηση της ισότητας λοιπόν μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να εξετάσουμε με περισσότερες ε, λεπτομέρειες και με περισσότερη προσοχή τον προϋπολογισμό. Να υπάρχουν ε, περισσότερες υψηλόβαθμες δεσμεύσεις στην ε, ισότητα των φύλων διότι, ενακολουθήσουμε τη ροή του χρήματος, θα δούμε πόσο ο προπολογισμό ε, αντανακλά αυτές τις ε, υψηλόβαθμες ε, αποφάσεις. Αυτό φαίνεται στο πώς δαπανώνται κονδύλια. Σκοπός λοιπόν είναι η βελτίωση της λογοδοσίας και η βελτίωση της ισότητας των φίλων σε όλους τους τομείς του προπολογισμού. Επίσης, αναμένουμε να βελτιωθεί και η υποβολή ε, εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο για την ισότητα στον προπολογισμό και να ε, βελτιωθούν οι πολιτικές. Έτσι λοιπόν η συνεκτίμηση της ισότητας των φίλων στον προϋπολογισμό μας δίνει ένα σημείο αναφοράς, μας δίνει ένα σημείο παρέμβασης έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο διάφορων στόχων όπως η ισότητα των φίλων και συνεκτίμηση της διάστασης του φίλου. Αυτή λοιπόν ε, η μέθοδος είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που βοηθά στην βελτίωση της δημοκρατικής λογοδοσίας στον προπολογισμό. Κατά την πιλωτική μας ε, μελέτη λοιπόν βασιστήκαμε σε μία στιβαρή μεθοδολογία ε, που προσεγγίζει τις δυνατότητες που έχουμε προσπαθούμε να αξιολογήσουμε διάφορες στοιχεία του προπολογισμού για να δούμε πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζουν το θέμα της ισότητας ε, ως προς την κατανομή των πόρων και την ε, χρήση τους. Χρησιμοποιούμε την ε, μέθοδο του να υιοθετούμε μια εξωτερική προσέγγιση. Βλέπουμε τους ε, ποιους στόχους ε, προβλέπουν οι συνθήκες και πώς ε, αυτοί επιτυγχάνονται. Προσπαθούμε να δούμε τα μέτρα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, που εισαγάγονται στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μετρηθεί η πρόοδος αυτών με βάση εξωτερικών συγκριτικών μεθόδων. Στη μελέτη, επίσης, προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ισότητα έχει επιπτώσει σε διάφορους τίτλους του προϋπολογισμού. Έχουμε εφαρμόσει την μεθοδολογία και ε, προσπαθούμε να δείξουμε τα αποτελέσματα αυτής. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας ε, για να δούμε εάν εσείς θεωρείτε την μέθοδο που ακολουθήσαμε χρήσιμη. Διεξήγαμε την ε, έρευνα αυτή σε διάφορους τίτλους του προπολογισμού και διαπιστώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις λείπουν στατιστικά στοιχεία μας, λείπουν πληροφορίες που καθιστούν δύσκολο το έργο μας. Είναι ένας μεγάλος περιορισμός ε, και θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στις ε, ελλείψεις αυτές. Εάν θέλουμε να αυξηθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η λογοδοσία στον προπολογισμό, τότε χρειάζεται να καλυφθούν αυτά τα κενά στις πληροφορίες και στα στατιστικά στοιχεία, έτσι ώστε να βοηθήσει αυτό στο έργο μα. Χρειάζονται λοιπόν βελτιώσει στη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού έτσι ώστε να συνεκτιμηθεί η ισότητα των φύλων και να βελτιωθεί και η όλη διαδικασία στο μέλλον. Υπάρχουν ε, διάφορε συστάσει που έχουμε ε, κάνει έτσι ώστε να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική και δημοσιονομική ε, λογοδοσία. Και στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου κυρία Συγκάς. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σα δώσω μερικέ ε, επιπλέον πληροφορίε για την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και τα κύρια ευρήματά μα. Υπάρχει και ένα παράρτημα στην μελέτη μα όπου εξηγείται με λεπτομέρειε η μέθοδος που ακολουθήσαμε και θα βρείτε στην σελίδα 16 αυτό το παράρτημα. Όπω είπε και η Φιώνα, εμεί ακολουθήσαμε μια προσέγγιση βασισμένη στις δυνατότητες, ανθρωποκεντρική, ουμανιστική αν θέλετε προσέγγιση, και εστιάσαμε όχι τόσο στα ποσά και στα χρήματα, αλλά σε συγκεκριμένες δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής άνδρων και γυναικών και είδαμε σε ποια έκταση τόσο άνδρες όσο και γυναίκες έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δραστηριότητες. Αποφασίσα, καταλήξαμε λοιπόν σε πέντε κύριες δραστηριότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ βασικές για να ε, εκπληρώνεται η επιθυμητή ποιότητα ζωής. Ισότητα στην εργασία, ισότητα στην ε, οικογένεια, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην συμμετοχή στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στο πολιτικό σύστημα, στην ε, ε, έκφραση πολιτικών απόψεων, έκφραση ε, αυτοδιάθεση, ίση πρόσβαση σε ε, αρμονική διαβίωση, ίση πρόσβαση σε καταφύγια, ε, ισότητα στην προσωπικότητα, ίση πρόσβαση στην ανάπτυξη διάφορων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, στην πνευματικότητα, στις θρησκευτικές δραστηριότητες, στις σωματικές ε, δραστηριότητες, απόλυτη ισότητα και έλλειψη παραγόντων ε, εκφοβισμού. Εξετάσαμε λοιπόν όλους αυτούς τους παράγοντες που για μας ε, κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ποιοτική και πιο εύκολη και είδαμε πώς αυτές οι πτυχές αντικατοπτρίζονται στον προπολογισμό και προσπαθήσαμε να δούμε ποιες ικανότητες θα έχουν επιπτώσεις στην πραγματική ζωή και ε, ποια, θα είναι, ποια θα είναι η έκταση αυτών των επιπτώσεων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τους τίτλους του προπολογισμού και ποιοι από αυτούς αντανακλούν την πραγματική ισότητα. Είδαμε λοιπόν ότι όσο υψηλότερο το όσο ψηλότερος ο αριθμός και ένταση των ικανοτήτων, τόσο μεγαλύτερη και η επιρροή στον ε, προπολογισμό και στην ε, πολιτική αυτού. Κοιτάξαμε επίσης ε, τις δαπάνε και τις αποφάσεις για τις δαπάνες για να δούμε εάν έχει ληφθεί υπόψη η ισότητα των φύλων. Μετά διαπιστώσαμε ότι με εξετάζοντας αυτά μπορούμε να καταλάβουμε εάν έχει συνεκτιμηθεί η διάσταση της ισότητας στην διαδικασία κατάρτισης σε προπολογισμού. Κοιτάξαμε επίσης και, την, και το στάδιο της εφαρμογής, τους δικαιούχους και προσπαθήσαμε να δούμε πόσο έχουν επωφεληθεί άνδρες και γυναίκες και αν ε, έχουν επωφεληθεί με ίσο τρόπο. Τέλος, προτείναμε κάποιες ε, δράσεις. Προτείναμε καταρχάς μία επανεξέταση και αξιολόγηση των εφιστάμενων δράσεων και βελτίωση αυτών. Η δομή έχει ω εξή. Όπως βλέπετε και στην διαφάνεια υπάρχει μια ανάλυση. Έχουμε καταρχάς το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους και διάφορα, διάφορα άλλα ταμεία και δομές που δίνουν τη δυνατότητα ε, ισότητας, πρόσβαση στην ισότητα. Κοιτάξαμε επίσης τις διάφορες ε, δυνατότητες που δίδονται στους, ε, ε, στις ομάδες, στις λιγότερο... Στις ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τις δυνατότητες που έχουν για ένταξη στην κοινωνία, κοιτάξαμε τις περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικού αποκλεισμού, αναλύσαμε τα κοινωνικο-οικονομικά και οικονομικοπολιτικά συστήματα, την αγορά εργασίας και την πρόσβαση, την ίση πρόσβαση σε αυτή. Και διαπιστώσαμε ότι ναι μεν υπάρχει ο στόχος της ισότητας σε γενικότερη έννοια και σε υψηλό επίπεδο, όμως δεν διαφαίνεται παντού σε κάθε πτυχή του προϋπολογισμού και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ως προς την εφαρμογή, για παράδειγμα της ίσης κατανομής επόρων, της εφαρμογής σε μεθόδων που θα οδηγήσουν σε αυτήν την συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων. Μετά, η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν συγκεκριμένη διότι είχαμε και συγκεκριμένους χρονικούς και οικονομικούς ε, περιορισμούς. Πιστεύουμε πως ε, πρέπει να είναι οριζόντια η ε, μεθοδολογία και οριζόντια εφαρμογή της συνεκτίμησης της ισότητας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, διότι είναι και οριζόντιο το ζήτημα. Θα έχει άμεσα και πιο ορατά ωφέλει μια οριζόντια εφαρμογή. Διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε από το να χρησιμοποιηθεί σε επιλεκτικούς, ε, σε επιλεγμένους τομείς η διαδικασία της συνεκτίμησης της ισότητας. Τώρα, ας δούμε κάποια συγκεκριμένα νούμερα. κράτη-μέλη τα οποία έχουν χαμηλές ε, αναλήψεις υποχρεώσεων για την συνεκτίμηση της ισότητας θα μπορούσαν να κάνουν διάφορες δράσεις για να βελτιώσουν αυτό το θέμα. Θα σας δώσω κάποια θετικά και κάποια αρνητικά παραδείγματα για την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και της ε, βιομηχανοποίησης υπάρχει περιθώριο ε, βελτίωση της ίσης εκπροσώπησης των ανδρών και γυναικών στις ε, στον βιομηχανικό κλάδο. Και εδώ χρειάζεται η ισότητα των φύλων να μπει ε, στο, στην ατζέντα των εργοδοτών, των εργοδοτών στον κλάδο της βιομηχανίας. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει, διότι η ισότητα των φύλων δεν αναγνωρίζεται ως στόχος πολιτικής στην βιομηχανία. Ένα θετικό από την άλλη παράδειγμα είναι ε, ορίζοντας 2020. Υπάρχουν ισχυροί στόχοι ισότητας ε, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, ιδιαίτερα στους ε, τομείς, στον τομέα της εκπαίδευσης και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχει επίσης και ισχυρότερη ευρωπαϊκή δέσμευση για μακροπρόθεσμη βελτίωση της ισότητας στον ε, χώρο της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Τώρα, ένα άλλο αρνητικό παράδειγμα είναι κλάδι όπως ε, τα μέσα ενημέρωσης, οπτικό-ακουστική βιομηχανία. Εκεί βλέπουμε πως υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, ιδιαίτερα σε υψηλόβαθμες θέσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Εδώ πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία για μια θετική αλλαγή. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τα πράγματα και να θέσει ως ε, στόχο προτεραιότητα σε την πολιτική ισότητα σε αυτούς τους χώρους. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί αυτό γρήγορα, διότι μέχρι τώρα ούτε σε αυτόν τον τομέα έχει αναγνωριστεί η ισότητα ως ε, κύριος στόχος πολιτικής. Τώρα, ποια είναι τα κύρια ευρήματά μας. Καταρχάς, Στι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Χάρτα των Αθεμελιωδών Δικαιωμάτων υπάρχει μεν υψηλόβαθμη δέσμευση για την ισότητα των φύλων, όμω όσο προχωράμε προς τα κάτω, όσο καταβαίνουμε επίπεδα και φτάνουμε στην εφαρμογή της πολιτικής, βλέπουμε ότι δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν έχει υλοποιηθεί από την βάση. Για παράδειγμα, σε τίτλους του προπολογισμού που ασχολούνται με εσωτερικά θέματα και θέματα δικαιοσύνης βλέπουμε πως ε, οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής επισκιάζουν τους στόχους ισότητας. Τώρα, όσον αφορά την απασχόληση, την ε, εκπαίδευση και την, ε, την κοινωνική συμμετοχή, είναι λίγο βελτιωμένα τα πράγματα εκεί, όμως το πρόβλημα παραμένει. Διότι τι γίνεται, υπάρχουν διάφορες... υπάρχουν διαφορές μάλλον στους επιμέρου τομεί. Σε κάποιου τομεί αναγνωρίζεται ισότητα ως κύριος στόχο προτεραιότητας, σε κάποιους καθόλου. Και ιδιαίτερα μάλιστα μετά την οικονομική κρίση βλέπουμε ότι τα θέματα ισότητας ε, είναι διασυνοριακά και οριζόντια. Ε, υπάρχουν, υπάρχει φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστευση, σεξουαλική ε, βία και αυτά τα θέματα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο με συγκεκριμένες δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωριστεί η ισότητα των φύλων ως ε, κύριος στόχος. Διαφορετικά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη βάση. Αλλά βασικά ευρήματα είναι ότι οι τίτλοι του προϋπολογισμού πολλές φορές δεν έχουν αρκετή διαφάνεια, είτε ως προς τα ποσά που ε, κατανέμονται για την ισότητα, είτε για παράδειγμα στο τομέα της δικαιοσύνης είδαμε πως υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία προσπαθούν με να επιτύχουν στόχους πολιτικής ε, στα, στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπάρχουν και κάποια προγράμματα με, που εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα κατά πολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Βλέπουμε όμως ότι Τώρα αυτές, αυτοί έχουν ε, συγχωνευθεί, αυτή η τίτλη προπολογισμού και δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε τι συμβαίνει, ποιοι είναι οι επιμέρους ε, στόχοι. Και εδώ επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να επισκιάσουν ε, άλλοι στόχοι την ισότητα. Επίσης, ε, δεν γίνεται σαφής ε, διαχωρισμός ε, των ομάδων στις οποίες στοχεύουν αυτές οι πολιτικές. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη διαφάνειας και εκεί, αλλά και σε θέματα χρηματοδότησης. Πρέπει να δούμε Ποιε είναι οι, οι κύριες ομάδες τις οποίες πρέπει να εστιάσουμε τις ε, δαπάνε μας. Όσο δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε εντοπίσει αυτές ε, τις ομάδες, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να περάσουμε στο στάδιο της εφαρμογής και να δούμε μετά εάν έχουν υλοποιηθεί αυτοί οι στόχοι και εάν οι ε, δικαιούχοι έχουν όντως αποκομίσει τα ωφέλη της πολιτικής μας. Και τώρα θα δώσω το λόγο πάλι στη Φιώνα, η οποία θα σας ε, αναφέρει τις συστάσεις μας. Για να συνοψίσω λοιπόν γρήγορα γρήγορα. Πρώτη υπόδειξη. Πιστεύω ότι θα πρέπει η ισότητα των φίλων να αναγνωριστεί ως στόχος πολιτικής σε όλους ε, τους τίτλους του προϋπολογισμού και θα πρέπει το gender mainstream να συμπεριληφθεί επίσης στην υλοποίηση των πολιτικών. Θα πρέπει επίσης ε, ε, συγκεκριμένα ποσά να διατεθούν για δράσεις που θα πρέπει να αναφέρονται στον προεπολισμό συγκεκριμένα για αύξηση της διαφάνειας, γιατί πολλοί λόγος έγινε και το πρωί για την ανάγκη διαφάνειας στον προεπολεξμό. Και επίσης συγκεκριμένοι δείκτες ε, και δεδομένα για την ισότητα των φύλων που θα πρέπει να συλλέγονται και να δημοσιεύονται σε τακτά διαστήματα. Τώρα για το ρόλο τη δική σας επιτροπή ή άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου και άλλων ενδιαφερομένων, τι ρόλο μπορούν να έχουν. Ε, για να έχουμε μια επιτυχημένη διαδικασία συνεκτίμησης τη διάσταση των στον προπολογισμό σημαίνει ότι όλα τα όργανα τη Ένωση και όλοι οι φορεί, όλοι οι εκτελεστικοί οργανισμοί θα πρέπει να μπορούν του δείκτε και τι ομάδε στόχο σε σχέση με τους άτομα να μπορούν να τα χρησιμοποιούν όταν ζητούν χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιούνται οι κατευθυντήριε γραμμέ και να είναι και παρκώ διαφανέ το σχέδιο προπολογισμού. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει στο πλαίσιο τη διαδικασία κατάρτιση, έγκριση του προπολογισμού και χορήγηση απαλλαγή να εξασφαλίσει τη λογοδοσία σε ό,τι αφορά ε, την τήρηση αυτή τη διαδικασία για την ισότητα των φύλων και την εκτίμησή τη. Ολοκληρώθηκε εδώ η παρουσίαση. Θα θέλαμε να μα πείτε πόσο χρήσιμη θεωρήσατε τη μεθοδολογία ε, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αδυναμιών στι πολιτικέ για την ισότητα των φύλων, πόσο αποτελεσματικά μπορούν να αντιμετωπιστούν οι βασικέ προκλήσει. Μπορούμε να έχουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά την παροχή πιο αναλυτικών πληροφοριών, πλήρω κάποιων κενών πληροφόρηση, πιο διαφανή προπολογισμό ώστε να μπορούν καλύτερα ε, να παρακολουθούνται οι στόχοι το πώς εφαρμόζονται. Και αυτό το μοντέλο του gender budgeting ε, συνιστά μια προστιθέμενη αξία ε, και για εσάς και για όσους επιθυμούν να υπάρχει καλύτερη λογοδοσία στα θέματα ισότητας των φίλων στην Ένωση και στις πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Merci, pour... Euh, Κυρίες μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αλλά πρέπει να σας πω ότι η γραμματεία της Επιτροπής Προπολογισμών δεν σέβεται την ισότητα των φίλων Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία γυναικών, οι οποίες ασκούν και μια εξουσία πάρα πολύ βέβαια θετική, την οποία αναγνωρίζω, αναγνωρίζουμε, γι' αυτό δώσω το λόγο και στην Πατρίσια Σουλίν, ευθύ αμέσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζω τη μελέτη αυτή για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή και την εισόδο των φίλων και να ευχαριστήσω του συναδέλφου και τις συναδέλφου από την Επιτροπή ΦΑΜ που έλαβαν την πρωτοβουλία για τη μελέτη αυτή και να ευχαριστήσω όλου σα ε, για την παρουσίαση αυτή τη εκθέσης σήμερα και ευχαριστούμε και για τι συστάσει σα. Για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι χρειαζόμαστε πολιτική και οικονομική όμω στήριξη. Γι' αυτό συζητήσαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε να συζητάμε πιστεύω ε, για αυτή την οικονομική στήριξη που προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ένα ισχυρό εργαλείο υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θα ήθελα επίσης ε, να επισημάνω ότι εδώ και πολλά χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για την ισότητα των φύλων. Πρόκειται για έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την πλήρη μας στήριξη. Όπω είπε ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πολιτικής του κατευθυντήρε γραμμέ, και παραθέτω τώρα είπε η ισότητα των φίλων δεν είναι πολυτέλεια είναι πολιτική αναγκαιότητα φυσικά διαρκώ διερωτώμεθα κατά πόσο αυτή η πολιτική στήριξη είναι αρκετή ή αν έχουμε μείνει πίσω ε, τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάσατε είναι πιστεύω διαφωτιστικά για όλους μας ε, δείχνουν ότι η οικονομική στήριξη για την ισότητα των φύλων και ειδικά η στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες ε, βάσει της πολύ καλά τεκμηριωμένης και παρουσιασμένης μελέτης αυτής. Επιπλέον η όλη διαδικασία δεν είναι απόλυτα διαφανής, δεν είναι σαφές πόσα χρήματα δαπανώνται για συγκεκριμένους στόχους και μέτρα. Και οι δείκτες ε, των φύλων δεν παρακολουθούνται ούτε χρησιμοποιούνται αρκετά συστηματικά ώστε να αξιολογούν επαρκώς την αποτελεσματικότητα των επιμέρους μέτρων. Φυσικά δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας. Ε, καταβάλουμε προσπάθειες για βελτίωση των πραγμάτων και Ίσως βέβαια να θέλαμε τα αποτελέσματα να ήταν καλύτερα, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο για να βελτιώσουμε τη δόμηση του προπολογισμού στο μέλλον. Τέλος, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε. Ε, θα ήθελα να πάρει το λόγο όποιο θέλει να υποβάλει του στους μα. μας. Θα ήθελε κάποιο το λόγο. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Η μελέτη αυτή πιστεύω είναι πολύ διαφωτιστική. Ξέρετε, δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε όλα σε προπολογισμό. Η ισότητα των φίλων είναι αρχικά θέμα ηθικής και αξιών. Παρά τις προσπαθίες μας για διαφάνεια, δεν μπορούν να εμφανίζονται όλα στα ε, κονδυλία του προπολογισμού. Πρόκειται για επιπλέον ε, στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τη Διευθύνση Ανθρωπινών Πόρων. Ε, αυτή θα μπορούσε να μας διαφωτίσει, να μας δώσει δείκτες. Πρόκειται για ε, τους απολογισμούς ε, του τι συμβαίνει στην κοινωνία όλα αυτά είναι συμπληρωματικές πληροφορίες πέραν των προϋπολογισμών μας ε, εσείς κατά κάποιο τρόπο μας προκαλέσατε με, δημιουργώντας κάποια ερωτήματα η Πατρίσια Σέλεγη πιστεύω θα είναι ο θεματοφύλακας κατά τη διάρκεια των εργασιών μας ώστε να βεβαιωθεί ότι αυτή η αναφορά στην ισότητα των φύλων δεν θα παραμείνει στη θεωρία ότι θα είναι ένα ηθικό πρόσταγμα το οποίο εμείς ε, τηρούμε καθημερινά ε, προς εξυπηρέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε λοιπόν ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, χαιρόμαστε που σας είδαμε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον στο πλαίσιο αυτών των εργασιών. Ευχαριστούμε. Τα είπατε όλα μέσω της εξαιρετικής σας παρουσίασης. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. ευχαριστή και ο Πρόεδρος. Bien, mes chers collègues, Συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι τις εργασίες μας. Να σας αναφέρω ποιες ήταν οι αποφάσεις ε, χθες των συντονιστών. Δύο τον αριθμό. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και Ταμείο Λυγγύη. Ήταν ε, οι δύο φάκελοι που επελέγησαν για το διάλογο που έχουμε οι συγητές των ε, επιτροπών των αρμόδιων και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο νομοθετική διαδικασία, διαδικασίας. Επόμενη stakeholders, δεύτερη απόφαση, η ΕΕΔ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, θα κληθεί κατά εφαρμογή του άρθρου 123 του καθεστώτο που εφαρμόζει του λοιπού ε, στα λοιπά όργανα τη Ένωση για ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πρόθεσή τη να ορίσει ειδικό σύμβουλο. Αυτό θα λάβει χώρα στην επόμενη συνεδρία σε σε Προϋπολισμών. Ειδικό σύμβουλο ε, για συνέδρια και συγκεκριμένα με στόχο την ειρήνευση στην Κολομβία. Αυτές είναι οι δύο αποφάσεις που έλειψαν χθες συνεδρίες των συντονιστών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον συνάδελφο Χριστοφόρου, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την πληρωμή προκαταβάσεων στο πλαίσιο του 2016. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ε, απόφαση του και την πρότασή του μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντα υπόψη τόσο την έκθεση τη Επιτροπή τη Δευτέρα Δεκεμβρίου του 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη Επιτροπή, αλλά και την τροποποίηση που εμεί ήδη ένθερμα υποστηρίξαμε ω Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά την δυνατότητα να εκταμιεύεται 10% ποσών ω προκαταβολή για την στήριξη όλων εκείνων οι οποίοι πλήττονται από φυσικέ καταστροφέ, θεωρώ ότι ο στόχο του Ταμείου, όπου ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά άμεσα αποτελεσματικά και με ταχύτατο τρόπο, προσφέροντα το μάξιμο μέχρι και 10% του ποσού του Ταμείου και τη αποζημίωση ω προκαταβολή σε πληγέντε από φυσικέ καταστροφέ, πιστεύω είναι στόχο προ την ορθή κατεύθυνση, γιατί ουσιαστικά και εμεί μέσα από αυτή την Επιτροπή πολλές φορές τονίσαμε τη γραφειοκρατία, τις διαδικασίες και για το άλλα ταμεία κινητοποιήσεως που αφορούσαν την παγκοσμιοποίηση που ουσιαστικά οι βοήθειες φτάνουν πολύ αργά στους κατοίκους και στις πληγήσεις περιοχές αλλά πολύ περισσότερο με αυτή την αμεσότητα θα μπορούμε να ανακουφίσουμε όλους εκείνους οι οποίοι πλήττονται και αναμένουν να ολοκληρωθούν ατέρμονε διαδικασίε για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα ε, προ αυτή την κατεύθυνση. Το ποσό, το ανώτατο, το μέγιστο ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια, άρα από αυτά μάξιμο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 50 εκατομμύρια ω προκαταβολή. Είναι σημαντικό δεν να αναφέρω ότι αυτά τα οποία θα δίνονται ω προκαταβολή, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να τα επιστρέψουν μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της χρηστής διαχείρισης. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή την έκθεση και μέσα από αυτή την ψήφιση στέλνουμε ένα ξεκάθαρο, σαφέστατο μήνυμα ότι τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να γίνονται πραγματικά όχι ταμεία γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά ταμεία που επιδεικνύουν αλληλεγγύη και άμεσα φτάνουν εκεί που πλήττονται περιοχέ είτε από φυσικέ καταστροφέ είτε για άλλου λόγου στου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο πολύ πολλέ φορέ τα έχουν ανάγκη και βρίσκονται σε απόγνωση αναμένοντα πότε θα φτάσουν τελικά τα χρήματα για να υπάρξει αυτή η ανακούφιση αλλά και αυτή η έμπρακτη συμπαράσταση. Και μπορώ να τονίσω ολοκληρώνοντα ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το να καταβάλουμε την προκαταβολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τόσο άμεσα και τόσο κοντά στους πολίτες που έχουν ανάγκη και που πλήττονται από διάφορες φυσικές καταστροφές και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να καταστεί και έναν καλό παράδειγμα για τη λειτουργία και των άλλων ταμείων που χρησιμοποιούμε ε, ω Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά από αυτά τα ταμεία του προπολογισμού του εξετάζουμε και εμεί ω Επιτροπή που δυστυχώ οι βοήθειε αυτέ φτάνουν πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα και σίγουρα και η αποτελεσματικότητα αυτών των χρημάτων μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Merci, monsieur le rapporteur. Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα όλα είναι απολύτως σαφή. Να σας αναφέρω ότι η κατάσταση των τροπολογιών θα πρέπει να γίνει ε, το αργότερο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου ώρα 12 το μεσημέρι και σε ό,τι αφορά ε, την ψηφοφορία δεν έχει ακόμη προβλεφθεί ημερομηνία. Ούτε στην Επιτροπή Προπολογισμών, ούτε βέβαια και για την Ολομέλεια. Τώρα, ερχόμαστε στο ψήφισμα για το σχέδιο προπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 ε, να επαληθεύσουμε ε, για πέντε λεπτά προτείνω να διακόψουμε για να επαληθεύσουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Oui, pour Profitez-en ε, Μπορείτε να αποφεληθείτε του διαλύματος για να βάλετε στο μηχάνημα που είναι μπροστά σας τις κάρτες. Ah oui, alors. Ψηφοφορία έχει προβληθεί για τις 11, ακούστηκε. Λοιπόν, κανονικά λέει ο πρόεδρος, ε, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε πριν τις 11. Οπότε αναστέλλονται οι εργασίες μας μέχρι τις 11.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 το βέβαια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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE La séance est reprise. Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση και τώρα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για το ψήφισμα επί του πολιτικού μηνύματος ε, που βασίζεται στις ψηφοφορίες μας 28 ε, και 29 Σεπτεμβρίου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016. Το ψήφισμα αυτό έχει ως συζητητές τον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες και τον Ζεράρ Ντεπρέ. Να σας ζητήσω να, παρουσ... να βάλετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες στις συσκευές ώστε να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, δεν λειτουργεί όμω. Τι συμβαίνει. Δεν υπάρχουν συσκευέ για τι κάρτε. Δεν υπάρχει συσκευή ψηφοφορία λέμε. Θα ψηφίσουμε διανατάσεις χειρός. Δεν υπάρχουν μηχανηματάκια. Γιατί. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, μέχρι να λύσουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα, να δώσω τον λόγο στους γενικούς ηγητές, διότι στις ψηφοφορίες 25 29 Σεπτεμβρίου δεν φάνηκε μετά από εξέταση ότι υπήρχαν κάποιες προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν, οι οποίες ε, είχαν διαφύγει παρά την ε, επιμελή επανεξέταση του κειμένου. Οπότε πρέπει να προβούμε σε απαραίτητε διορθώσει και για αυτόν τον σκοπό δίνω τον λόγο στον Χωσέ Μανώλη Φερνάντε, το έγγραφο που έχετε μπροστά σα. Κύριε Γενικέ Εισηγητή, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για συνήθειε διορθώσει ε, και προσαρμογές ε, τεχνικής φύσης αντί να γίνουν στην Ολομέλεια καλύτερα να γίνουν ήδη εδώ τώρα και όπως είπα είναι κάτι που συνηθίζεται είναι απλά τεχνική φύσης λοιπόν για την επικεφαλίδα 1α στη γραμμή 04030201 στο παράρτημα της λίστας ψηφοφοριών δεύτερο υπομπλοκ above DB η, το, η λάθος λέξη είναι το λάθος ποσό είναι 3.594 ευρώ αντί για 3.954. 5.94 λοιπόν αντί για 9.54. κάποιο αντέστρεψε ψεύτιμος κατά Το σωστό ποσό λοιπόν είναι 3.594.000 ευρώ. Στην επικεφαλίδα 4, πληρωμές γραμμή 22040103 στη λίστα ψηφοφορία για τι πληρωμέ δεύτερο, ε, δευτερεύον μπλοκ ε, από DB. Τα ποσά προσέχθηκαν δεν ευθυγραμμίζονται με τη συμφωνημένη στρατηγική για τι πληρωμέ ούτε με το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών ε, για τι δεσμεύσει. Πρέπει λοιπόν το ποσό να είναι. το ποσό πρέπει να είναι 10.200.000 ευρώ το σωστό ποσό της τροπολογιαστού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είναι 31.200.000 ευρώ αντί για 49.533.333 με τελικό ποσό 68.200.000 ευρώ για τα πιλωτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις στην επικεφαλήτα 2 γραμμή 0702-7728 για το TTIP για να ε, μην είναι χαμηλότερο το ποσό που έχει υιοθετήσει το Κοινοβούλιο από αυτό που προτείνει η Κομισιόν πρέπει να ανέρχεται σε 120.000 ευρώ. Στην νέα προπαρασκευαστική δράση, επικεφαλήτα 3, γραμμή 3302-7712 όσον αφορά την ένταξη των Ρώμα για να μην υπερβούν ε, οι πληρωμές ε, της αναλήψης υποχρεώσεων το ποσό πρέπει να ανέχεται σε 500.000 ευρώ Στην Επικεφαλή 5 γραμμή χ01021104 στη λίστα ψηφοφοριών για το τμήμα 3 διοικητικές δαπάνες η τροπολογία ΙΤΑ που υιοθετήθηκε ενισχύει την οριζόντια γραμμή χ01021104 κατά 40.000 ευρώ. Δεδομένη τη αιτιολόγηση αυτή τη τροπολογία και του συντάκτη της μπορεί να εξηγηθεί ότι η γραμμή προορισμού για αυτή την ενίσχυση πρέπει να είναι η 20.01.02.11. στο, κεφάλαιο, στο εμπορικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτές είναι οι προσαρμογές και οι διευκρινήσεις τεχνικής φύσης. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ Συγητή. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι. Ψηφίζουμε τις τροποποιήσεις αυτές, τροπολογίες αυτές με ναι, ανάθεση χειρός. Παρακαλώ. Ποιο συγκρίνει. Ευχαριστώ κατά. Δεν βλέπω αποχές. Δεν ναι, ναι, υπάρχουν αποχές. Μία αποχή. Εξακολουθεί να μην λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Μα τι συμβαίνει. Ε, σίγουρα θα ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρο, φυσικά, αλλά σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να μα δημιουργήσει πρόβλημα, θα χάσουμε χρόνο. Le premier amendement. Πρώτη τροπολογία. Αναβάλλεται για το τέλο ψηφοφορία. Στην παράγραφο. Πρώτη παράγραφο, τροπολογία 2 ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο 1, τροπολογία 3. Με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Ψηφίζουμε την τροπολογία, την προφορική. Ψήφι περ. Κατά. Ουδής. Αποχές. Όχι. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 2 τροπολογία 8 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία υπερθμών 9 όπου έχουμε και προφορική τροπολογία που θα τεθεί σε ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα από το recalls μέχρι και το regulation. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Μήπως πρέπει να ξαναμετρήσουμε. Όχι. Εγκρίνεται. Όχι. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Και, και θα μετρήσουμε. 14. ψήφοι κατά τώρα. 15 κατά. 14 υπέρ ήταν. Και πόσες αποχές έχουμε. Καμία. Μία. Άρα απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Όπως τροποποιήθηκε λοιπόν δηλαδή με τη συμπλήρωση του πρώτου τμήματος προφορικής, ψηφίζουμε α, μόλις άρχισε να δουλεύει το σύστημα. Άρα θα πρότεινα να βάλετε τις κάρτες για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία καταρχάς. Άρχεται η ψηφοφορία. 32 πρέπει να είναι οι ψηφίζοντες κανονικά. Κάποιοι περιμένουν. Δύο λείπουν. Ποιος δεν έχει ψηφίσει, ποιος δεν θέλει να ψηφίσει. Ενώ έχει βάλει την κάρτα του. Εντάξει, τώρα και τον κύριο Τάρν τον έχουμε υπόψη μας, δεν έχει την κάρτα του. Άρα η ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα τροπολογία 9. Όπως τροποποιήθηκε, συν το πρώτο μέσο προφορικής. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Άρα, η τροπολογία εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε. Τροπολογία 10. Στην παράγραφο 3, τροπολογία 10. Κύριε Πρόεδρε, κάποιος Συγγνώμη, νομίζω πως δεν ήταν αρκετά σαφές το τι ψηφίσαμε. Μας αφήσατε να ξαναψηφίσουμε την τροπολογία 9, την προφορική τροπολογία ή και τα δύο. Όλα μαζί. Τροπολογία 9, συν το πρώτο τμήμα της προφορικής τροπολογίας που είχε εγκριθεί. Το πρώτο τμήμα είχε εγκριθεί της προφορικής τροπολογίας. Άρα ψηφίσαμε την τροπολογία 9 όπως τροποποιήθηκε με συμπερίληψη του πρώτου τμήματος της προφορικής που είχε εγκριθεί προηγουμένως. Ωραία, σας παρακαλώ λοιπόν τότε να επαναληφθεί η ψηφοφορία, διότι κατά την καταμέτρηση είχαμε και μία ψήφο κατά. Και τώρα πιστεύω πως ε, πολλοί ψήφισαν υπέρ χωρίς να ξέρουν για, χωρίς να ξέρουν ότι ψηφίζουν την τροπολογία. Σας παρακαλώ να επαναλάβουμε. Bon, alors. Μάλιστα. Άρα, θα ψηφίσουμε... Α, μισό λεπτό. Η κυρία Γκαρδία Θάμπαλ. Συγγνώμη, αλλά δεν είχαμε τον επικαιροποιημένο κατάλογο ψηφοφορίας, ε, άρα δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, μπερδευτήκαμε. Ε, και θα έλεγα ότι καλό είναι να ξαναθέσετε σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία γιατί εμείς τελικά θα ψηφίζαμε υπέρ του δεύτερου τμήματος. Α, λέει ο μάλιστα. Εντάξει. Επομένω. τώρα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της προφορικής τροπολογίας από το Recalls μέχρι το Regulation. Με ονομαστική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της προφορικής τροπολογίας. Ποιοι όχι. Όχι, ποιοι είναι υπέρ. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν το πρώτο 19 ψήφι 10 κατά και 5 αποχές. Δεύτερο τμήμα της προφορικής τροπολογίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φοβορίες. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. 26 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Το σύνολο τώρα... Α, όχι. Εγκρίνεται το σύνολο. Παράγραφος 3, τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην 4α νέα Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 με προφορική τροπολογία, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 16 ψήφι υπέρ, 14 κατά, 3 αποχές. Τροπολογία 15 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 20 κατά μία αποχή. Στην παράγραφο 8, τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Με προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8α νέα παράγραφος. Τροπολογία 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Πάμε. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Με προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 11. Τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Βάθος 11 αλφανέα, τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ, α, καταπίπτει εφόσον εγκρίθηκε η 33. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη 16α νέα 38. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ 12 κατά 3 αποχές. Τροπολογία 39 ψηφιπέ. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Ψήφι υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος τροπολογία 63. Εδώ έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα στην προφορική τροπολογία πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 19 ψήφιους κατά και 15 υπέρ. Τώρα, όπως τροποποιήθηκε η τροπολογία 63 με το πρώτο τμήμα, την ψηφίζουμε την 63, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, η τροπολογία ή ούτως τροποποιηθεί στα τροπολογία 63 εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 5, ψήφι υπέρ. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά Θα ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα, 19 προς 13. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 5 παράγραφος 31 τροπολογία 70 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 71 υπάρχει και μια τεχνική σφίσος διόρθωση ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, περνάμε σε συμβιβαστική 6 Εδώ τι έχουμε, ένα δεύτερο τμήμα. Όχι. Τι συμβαστική έξι ψηφίζουμε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Υπέρ. Με και τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81 με προφορική τροπολογία. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ψήφι πέρα. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Στο Τσαϊκλού. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 19 υπέρ, 14 15 υπέρ, 19 κατά. Λοιπόν, ε, επόμενη τροπολογία, 83 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 84 τροπολογία με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 94, τροπολογία 117, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στα υπόλοιπα τμήματα. Παραγραφός 62, τροπολογία 91. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Le scrutin est clos. Πέρας ψηφοφορίας ε, εγκρίνεται 22 10. Παράγραφος 60 α νέα τροπολογία 90 και παράγραφος 63 τροπολογία 92 και 93 οι τροπολογίες αυτές ε, αφού υπερψηφίστηκε η 91 θέλουμε λοιπόν πρέπει να έχουμε αφού ψηφίσαμε υπέρ της 91 πρέπει να ψηφίσουμε αφού εγκρίθηκε η 91 πρέπει να ψηφίσουμε την 90 και την 92 Πρέπει να τις ψηφίσουμε 90 και 92 μαζί ψηφίσουμε λοιπόν για την 90 και 92. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. να ψηφίσω και εγώ λέει ο πρόεδρος μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. évidemment. Si je mettais ma carte, ce serait quand même beaucoup mieux. Le scrutin est clos. τη Εγκρίνονται 22 έναντι 10. Οι δύο αυτέ τροπολογίε. 90 και 92. Περνάμε παράγραφο 63, τροπολογία 93. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παραγράφος 66 β νέα τροπολογία 96 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Σκοτάκι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται η τροπολογία με 17 κατά 14 υπέρ 2 αποχές τροπολογία 97 παραγράφου αλφα νέας ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 98 και 99 ίδιες. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές. Να ζητήσω να ψηφίσουμε τις 98 και 99 με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 έναντι 5 και 5 αποχές. Παράγραφος 77, τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Υπέρ, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 100. Πέρας ψηφοφορίας 16 υπέρ 16 κατά και ο κ. Σταράν ψήφισε υπέρ οπότε εγκρίνεται Donc il est adopté. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρο. 101 υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 102 της παραγράφου 77 συ νέο προφορική τροπολογία και με προφορική τροπολογία του εισηγητού τροπολογία 102 υπέρ Παράγραφος 77 Παράγραφος 77 Συ Τροπολογία 102 Με προφορική τροπολογία του εισηγητή Ποιος είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την προφορική τροπολογία του εισηγητή και τροπολογία που δεν έγιναν δεκτές. Γι' αυτό ως προσθήκη θα ήθελα να ψηφίσουμε χωριστά την τροπολογία από το request for the Secretary General to present to the Bureau σχεδόν ολόκληρη δηλαδή την τροπολογία των σοσιαλιστών μέχρι Parliament Estimates for the Budget of the Financial Year 2017. Ουσιαστικά είναι η τροπολογία των σοσιαλιστών χωρίς το πρώτο τμήμα για να είναι και συμβατό με το ότι έχουμε ψηφίσει μέχρι τώρα. Πολύ ωραία, είναι σαφές. Κύριε Εμείς είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας. Ah, Η προφορική τροπολογία ψηφίστηκε προηγουμένως. Περιμένετε διότι, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σιγητή. Κύριε Πρόεδρε, όπως το εξήγησα εγώ, αφού ψηφίσαμε την προφορική τροπολογία, δεν μπορούμε να έχουμε εδώ κανονικά άλλο τμήμα πάλι προς ψήφιση. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν θα το συμπεριλάβουμε αυτό το κομμάτι προς ψήφιση και αν το συμπεριλάβουμε μπορεί να σε εξήγησε και τους λόγους. Ε, εγώ προσπάθησα να παραμείνω πιστός σε αυτά που έχουμε ήδη ορίσει για να ευαίσθητο θέμα τον Ιούλιο και που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια. Οπότε μπορούμε να το θέσουμε σε ψήφιση, αλλά θα ζητήσω να το καταψηφίσουμε για τους λόγους που μόλις ανέφερα. Alors, <coughs> la règle Λοιπόν, ο είναι ότι αν υπάρχουν τρία μέλη που αντιτίθενται στην ψηφοφορία της προφορικής τροπολογίας ψηφίστηκε η προφορική τροπολογία αλλά αυτή είναι άλλη τροπολογία Α, είναι ε, ξεχωριστή ψηφοφορία αλλά δηλαδή, θεωρούμε ότι η προφορική τροπολογία δεν καλύπτει το μέρος το οποίο μόλις ε, παρουσίασε η κυρία Γκάρδια Ζαμπάν και ότι υπό αυτές τις συνθήκες το κομμάτι αυτό της αρχικής τροπολογίας θα μπορούσε να ε, τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτό είναι. Αυτή η αρχή λοιπόν, ε, λοιπόν για αυτή την ψηφοφορία, ποιος, ποιος είναι υπέρ να τη θέσουμε σε, σε ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε δηλαδή την αρχή της, του αν θα ψηφίσουμε ή όχι. Οπότε με ονομαστική ε, ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Σκριτά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το αίτημα με 19 ψήφους έναντι 13. Περνάμε στη συμβιβαστική β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Παραγράφος. Κύριε Σίγητε. Εκτός μικροφώνου, κύριε ομιλητής. Αυτό που θα πω τώρα δεν είναι πολιτικό πρόβλημα μεταξύ ομάδων, είναι πρόβλημα πραγματικό. Η παράγραφος 77 και η τροπολογία 104, η τροπολογία 109 και η 110 που αποσκοπούν ε, στην ανάθεση νέων αποστολών στον εσωτερικό ελεγκτή. Εγώ πήγα να δω τον οικονομικό κανονισμό, το δημοσιονομικό κανονισμό και το κείμενο αποσκοπεί στην ανάθεση αποστολών στον εσωτερικό ελεγκτή υπό τον έλεγχο του Προεδρείου. Εγώ πήγα λοιπόν να δω τον κανονισμό, τους κανόνες εφαρμογής του οικονομικού κανονισμού που λένε ότι ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά με απόλυτη ανεξαρτησία, με απόλυτη αυτονομία στην άσκηση των ελέγχων. Δεν μπορεί να λαμβάνει καμία οδηγία. Πολλέ λοιπόν από αυτές τις τροπολογίες, τροπολογίες τις που μόλι ανέφερα ε, δίνουν οδηγίες στον εσωτερικό ελεγκτή. Οπότε ζητώ λόγο, μη συμβατότητα με τον δημοσιονομικό κανονισμό να μην στηρίξουμε το κομμάτι των τροπολογιών που αφορούν τις νέες αποστολές που προτιθέμεθα να αναθέσουμε στον ιστορικό ελεγκτή ή να θέσουμε υπό ευθύνη του Προεδρείου. Οι σχέσεις μεταξύ του Προεδρείου και του ιστορικού ελεγκτή ρυθμίζονται από το χάρτη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Οικονομικών Ελέγχων που εθετήθηκε από το Προεδρείο 24 ε, Φεβρουαρίου του 2014. Θεωρώ λοιπόν ότι σοφό θα ήταν να μην δεχθούμε αυτές τις τροπολογίες. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ένας ε, ελεκτής υπόκειται σε κάποιον ε, και σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει ε, κάποιες οδηγίες λογικά από το άτομο αυτό στο οποίο υπόκειται αν το αφεντικό λοιπόν δεν είναι εκεί ο ελεκτής μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα είναι ο ανώτερος στην ιεραρχία συγγνώμη ε, σύμφωνα με το κείμενο εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Ο εσωτερικό ελεγκτή είναι απόλυτα αυτόνομο. Δεν μπορεί να λαμβάνει καμία οδηγία. Τέλο. λοιπόν, τώρα είναι τα Ο κύριο Φερνάνδη. Δεν ξέρω εάν οι σοσιαλιστέ θέλουν να αποσύρουμε τι τροπολογίε, αλλά μετά από τι εξηγήσει που δόθηκαν, θεωρώ ότι οι τροπολογίε αυτέ δεν μπορούν καν να ψηφιστούν. Ε, δεν είναι αποδεκτές αυτό τείνουμε να πιστέψουμε λέει ο Πρόεδρος διότι δεν είναι αποδεκτές οι τροπολογίες εφόσον έρχονται σε αντίθεση με το δημοσιονομικό κανονισμό δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Λοιπόν, ακούστε, ε, Πρόεδρος, θα ψηφίσουμε. Η άποψη του ΣΥΓΙΤΗ διατυπώθηκε σαφώς, βασίστησε σε ένα κείμενο το οποίο πράγματι θα μπορούσε να καταλήξει στο παράδεκτο των τροπολογιών αυτών διότι έρχονται σε αντίθεση με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Κύριε Σιγητά, ε, επιμένω σε αυτό που είπα και διευκρινίζω ότι αυτό ισχύει για τις τροπολογίε 104, 109 και 110 διότι και οι τρεις ε, βασίζονται στην ίδια λογική. Λοιπόν, απαράδεκτο. Ποιο ε, αποφασίζει το απαράδεκτο, ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Επιτροπή ολόκληρη. Α, εγώ. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαράδεκτε. Ε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτέ, κυρία Καρδιά Ζαβόλη. Δύο πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά η άποψη είναι δική σα, σωστό αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το μη παραδεκτών των τροπολογιών, θα σα παρακαλούσα να είστε πιο συγκεκριμένος, διότι είμαι βέβαιο ότι πληρώ, έχουμε ψηφίσει πολλές τροπολογίε για τον προπολογισμό που θα έπρεπε να είχαν κριθεί με παραδεκτέ και δεν έγινε αυτό. Δεν θέλω να αμφισβητήσω ότι εσείς έχετε τη δυνατότητα να πείτε ότι μια τροπολογία είναι μη παραδεκτή, το είχα πει και στην προηγούμενη θητεία. Απλά θα σας παρακαλούσα να κοιτάμε με τα ίδια μάτια και με τα ίδια γυαλιά, αν θέλετε, όλες τις τροπολογίες. Πρόεδρος, ε, θα προσπαθήσω να ασκήσω το δύσκολο αυτό καθήκον ε, ως το το πιο αμερόληπτα για να άρω κάθε υποψία μεροληψίας. Ο πρόεδρος, κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είναι ένα επικίνδυνο επιχείρημα αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος ο, δημο, ο, ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι ξεκάθαρος, σαφέστατος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο ψήφισμα το οποίο αντιβαίνει στον δημοσιονομικό κανονισμό. Εν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά την ανεξαρτησία την οποία υποτίθεται πως έχουμε, τότε πρέπει να τη διασφαλίσουμε κιόλα. Δεν πρέπει να μπούμε σε τέτοιες ε, άλλες αρμοδιότητες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως θα ήταν καλύτερο εάν η ομάδα σας ε, δεν συνεχίσει αυτήν την ε, διαφωνία, αλλά να αποδεχτεί ότι το κείμενο πρέπει να είναι έτσι σαφές. Μιλάμε για το δημοσιονομικό κανονισμό. À Μήπως να αποσύρετε την τροπολογία σας, λέει ο Πρόεδρος. για να μην την κρίνω μη παραδεκτή δηλαδή. Λοιπόν, για να έχω ίσχυτη συνείδησή μου, θα θέσω σε ψηφοφορία την 104. Και αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δεν θα θέσω σε ψηφοφορία τις άλλες δύο, δηλαδή την 109 και την 110. Ένσταση. Ο κύριο Ντεπρέ, για το 104 εγώ λέω να τεθεί σε ψηφοφορία αλλά την τελευταία παράγραφο να μην την ψηφίσουμε. Αν θέλουμε να σεβαστούμε τη λογική που εγώ υπερασπίστηκα, θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας 104, άρα αυτό συνεπάγεται την διαγραφή της ε, αμφιλεγόμενης ε, φράσης «Considers that this overview should be validated by the internal auditors and responsibility of the Parliament's Bureau». Ψηφίζουμε τροπολογία 104 όπως διορθώθηκε από τον εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Donc, euh, Επομένως, η Επιτροπή Προπολογισμών θεωρεί πως δεν μπορεί το Προεδρείο να υποκαταστήσει τι αρμοδιότητε του ελεγκτή. Άρα 109 και 110 δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Τροπολογία 105, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται τροπολογία 107 με προφορική τροπολογία για διαγραφή του τμήματος An Open Dialogue and Should Ensure. Υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Ήταν 107. Έρχεται 108 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 και 10 δεν έχουν καταπέσει. 111 τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 καταπέ, έχει καταπέσει. Η κυρία Γκαρδιά Συγγνώμη που περιπλέκω τόσο πολύ τα πράγματα, ε, αλλά όπως ακριβώς ε, και πριν από κάποια ψηφοφορία είχαμε ζητήσει για μια προηγούμενη ψηφοφορία αυτό που θέλουμε να στήσουμε και για την 112, δηλαδή να ψηφιστεί ως προσθήκη να μην ε, καταπέσει. Γιατί ουσιαστικά μιλάει για τις γενικές δαπάνες και πως γίνεται η απόδοση λογαριασμού λοιπά. Θα έλεγα λοιπόν το 112 να ψηφιστεί, αλλά ως προσθήκη το 111. Ο πρόεδρος Όλοι 112 ή ένα τμήμα της μόνο. Ένα τμήμα, ένα τμήμα, λέει η κυρία ε, Γκουέρντια Θάμπαλ. Για να δω από το... Inter-Al and Annual Declaration. Payment proof, modality of random controls. Oh, oh. Monsieur rapport. Κύριε Σιγητά, κύριε Σιγητά, κύριε Πρόεδρε, το συστήσαμε διαμακρόν. Αν προβούμε σε μια αυστηρή στενή ερμηνεία μπορούμε να πούμε ότι με το 111 που έγινε δεκτό ε, καταπίπτει το 112. Αν αποφασίζουμε τώρα να θέσουμε σε ψηφοφόρες προσθήκη το 112 δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να καταψηφίσουμε διότι εισάγει ε, διευκρινήσεις που δεν είναι αποτέλεσμα συνένεσης ε, μεταξύ μας. Αν είχαμε καταλήξει συνένεση θα συμφωνούσα να παραμείνει 112. Δεν υπήρξε συνένεση όμως σε σχέση με το πώς θα πρέπει να οργανωθεί αυτός ο έλεγχος και γι' αυτό το λόγο παρακαλώ να μην ψηφιστεί, να μην υπερψηφίσουν οι συνάδελφοι αυτή την τροπολογία. Και εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή, διότι πιστεύω πως πλέον έχει αποσαφωνιστεί με το 111 το πώς πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι παραδεκτό, παραδεκτή τροπολογία, γι' αυτό λοιπόν ε, ζητώ να ψηφίσουμε έτσι ώστε να διαλευκάνουμε τα πράγματα. Αν μου επιτρέπετε, λέω ε, θα θέσω σε ψηφοφορία μόνο τις τρει τελευταίες γραμμές, το τελευταίο τμήμα δηλαδή αυτή τη τροπολογία. Ε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, είναι σαφέ. Τροπολογία 114, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρόπο 115. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε τροπολογία 1, την οποία είχα αναβάλει για το τέλος Ποιοι είναι υπέρ της για σένα, Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τις γνωμοδοτήσεις ε, των εξειδικευμένων επιτροπών. Έχετε αντίρρηση να ψηφίσουμε από κοινού όλες αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Η ε, κυρία Γκρέσλε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ε, που διακόπτω την ψηφοφορία, αλλά είμαι συντάκτρια της γνωμοδότης Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και βλέπω ότι ε, σχεδόν σε όλες τις παραγράφους υπάρχει το σχόλιο out of scope. Να μιλάμε για την διαδικασία κατάρτισης του προπολογισμού. Και θέλουμε να βελτιωθεί η διαχείριση των Το out of scope δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το βάλατε, να μου το εξηγήσετε. Ο Γενικός ηγητής έχει εκφράσει την άποψη αυτή. Άρα, ο κ. Φερνάντες θα αυτός πρέπει να δώσει την απάντηση. Για ποια σελίδα μιλάμε, για τη σελίδα 10. Κοντ. Η Κοντ ο Γενικός Συγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για, μια γνωμο... για ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα πρέπει να είναι συνεκτικό, δεν πρέπει να υπάρχουν επαναλήψεις. Χρειάζεται κάποια λογική να το διατρέχει και να είναι κατανοητό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου εδώ αναγράφεται αυτό το out of scope. Και εγώ δεν συμφωνώ λοιπόν με αυτές γιατί δεν συνάδει με την γενικότερη λογική του ψηφίσματος. Θέλω λοιπόν να έχουμε ένα πολύ συνεκτικό και λογικό κείμενο εναρμονισμένο με τα προηγούμενα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί και με τις τροπολογίες μας. εάν εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα, πρέπει να συμφωνεί και με τις ε, δημοσιονομικές τροπολογίες που έχουμε ήδη ψηφίσει. Και να συμφωνεί και με άλλες ε, δημοσιονομικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τη Γραμματεία για την πολύτιμη βοήθεια σε ένα πολύ δύσκολο έργο. παρότι συμφωνούμε με πολλές από αυτές τις ε, προτάσεις, δεν μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε όλες και ε, να οδηγηθούμε σε ένα συνονθήλευμα που δεν βγάζει νόημα. Θέλουμε λοιπόν ένα ευανάγνωστο, συνεκτικό και κατανοητό κείμενο που θα συμφωνεί και με τις δημοσιονομικές ετροπολογίες που έχουν ήδη εγκριθεί και θα τις αντικατοπτρίζει επίσης. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το κείμενο όσα έχει και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Γκρέσλε που μας απέστησε την προσοχή σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σας προσπάθησα να σας εξηγήσω γιατί βάλαμε out of scope σε ορισμένε τροπολογίες, παρότι εγώ συμφωνώ με αυτό. Η κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εγώ θεωρώ λυπηρό το ότι όλοι οι κόποι που έχουμε καταβάλει για την ε, διαφάνεια των δημοσιονομικών και για την ε, χρηματοοικονομική, μηχανική τέλο πάντων που θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, δεν καταφέρνουμε να κρατήσουμε αυτά τα 59 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που μας φεύγουν από τα χέρια, που διαραίουν. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως είναι πάρα πολύ λυπηρό και δεν, δεν είναι κάτι το οποίο, για το οποίο πρέπει να είναι αυτή η Επιτροπή περήφανη. Πιστεύω πως θα ήμασταν ισχυρότεροι εάν στηρίζαμε ο ένας τον άλλο, αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλά και δεν έχουμε οδηγηθεί πουθενά. Ευχαριστώ. Μα χάρη σε εσάς έχει πλέον ξεκινήσει αυτή η συζήτηση ο Γενικό Συγητή. Να σα δώσω μία επιπλέον πληροφορία. Νόμιζα ότι είναι ξεκάθαρο σε όλου και όλε οι συναδέλφου. Είναι ότι οι γνωμοδοτήσει των επιτροπών προσαρτώνται, επισυνάπτονται. Δεν πετάγονται έξω από το παράθυρο. Συγκαταλέγονται τελικά στο ψήφισμα, συνενώνονται με το υπόλοιπο σώμα του κειμένου. Ο πρόεδρος Σίγουρα ε, σε ό,τι αφορά την προβλεψιμότητα θα λάβουμε υπόψη μα ε, τις παρατηρήσεις και απόψεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Του, του λεχθέντος παραμένουμε όμως ε, στην άποψη και εκτίμηση του Γενικού Εισηγητή. Συμφωνείτε λοιπόν να ψηφίσουμε συνολικά μαζί τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών επιτροπών. Άρα ψηφίζουμε από κοινού τις γνωμοδοτήσεις δεν καλύπτονται από άλλε παραγράφου που δεν καλύπτονται από άλλε παραγράφου ή δεν είναι εκτό θέματο out of scope. Υπέρ. Κατά. Δει. Αποχέ. Κανεί. Εγκρίνονται. Τώρα, το σύνολο του ψηφίσματος, όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ. 7 κατά. 4 αποχές. χαρητήρια Στους εισηγητές και σε όλους και όλες εσάς. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι ολοκληρώσαμε. Ο κ. Μάνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω απλά ένα σχόλιο. Όταν ψηφίζαμε για του εσωτερικού ελεγκτέ, αν αυτό είναι κατά των δημοσιονομικών κανονών, τότε και κάποιοι άλλοι θεσμοί όπω η ΕΚΟΣΟΚ έχουν την ίδια διευθύνση που συζητήσαμε και εμεί για την ψηφοφορία, οπότε πρέπει να υπολοιθέψουμε αυτά που είπε ο διότι δεν μπορεί να είναι κατά των κανονών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρχουν άλλοι θεσμοί που ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Ωραία, λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα έχουμε, θυμηθείτε, μία έκτακτη συνεδρίαση Budget Libre 19 Οκτωβρίου του 2015 εδώ στις Βρυξέλλες και ότι 22 Οκτωβρίου θα κάνουμε μια άλλη συνεδρίαση την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε δυστυχώς δεδομένων των κρατήσεων για τις αίθουσες και των περιορισμών της διερμηνίας. Ξέρω ότι μία από τις ομάδες έχει διάσκεψη την επόμενη εβδομάδα και τα μέλη της δεν θα μπορούν να είναι παρόντα. Λυπάμαι. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε φτάσει στο τέρμα της συνεδρίασης. Να σας υπενθυμίσω ότι απόψε στις 7 έχουμε μεικτή επιτροπή για τις ακροάσεις των υποψηφίων του Steering Board του FC για τις θέσεις Managing Director και Deputy Managing Director. Γενικού Διευθυντή και Αναστολική Γενικού Διευθυντή.